Guten Abend. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung des Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στην απόψινή συνεδρίαση. Ξεκινώ με το σημείο 1, υιοθέτηση τη μέσα διάταξη. Δεν έχω ανακοινώσει, Υπό το 2 να πω ότι έχουμε τυπώσει και το Cont News. Περνούμε τώρα στο σημείο 3 πολιτική κυριότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα και τον ε, διορισμό του Γενικού Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περνούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έχουμε 129 τροπολογίε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι έτοιμε οι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ την προσοχή στο γεγονό ότι το ψήφισμα αυτό είναι, μπορεί να υπογραφεί και μπορεί αυτό να τεθεί γραπτός όταν ε, επιβεβαιωθεί το κείμενο. Θέλετε να πάρετε το λόγο, υπάρχουν αντιρρήσεις, έχετε τις κάρτες σας. Θα πρέπει να μας πείτε μετά. Οργανωθείτε παρακαλώ με τις κάρτες σας. Εντάξει, ας περάσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία. προτείνω να ξεκινήσουμε με τις συμβαστικές τροπολογίες. Και να είναι έτσι απλούστερα τα πράγματα μετά. Συμβαστική Α, υπέρ. Συμβαστική Α. New, new paragraph 12a. New 12a new. Νέα παράγραφος 12α. A In favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Στην αναθεωρημένη εκδοχή που έχει διαμοιραστεί ως ε, έχει συμφωνηθεί στην Επιτροπή των Σκιωδών. Νέα παράγραφος πριν από την παράγραφο 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C, παράγραφος 22, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουν υιοθετηθεί όλες οι συμβαστικές τροπολογίες, έτσι απλουστεύονται τα πράγματα. Ξεκινούμε με την τροπολογία 14, γιατί 13 ήταν η συμβαστική Β. 14 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Το δεύτερο τμήμα αποσύρεται. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 και 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 25. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 28. Check is open. Check is over, and it is adopted. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 με προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 36. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 42. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά τη 43. Check And it is adopted. 44. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 56 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει. Το πρώτο τμήμα της 66. Πέρας. Ποιος άλλος δεν έχει κάρτα. Γιατί και εγώ ήθελα να ψηφίσω υπέρ. Έχετε την κάρτα σας, εντάξει. Εσείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσανέτσκι. Απορρίπτεται. 66. Yeah, yeah. 64 was in favor. 64 in favor. 60. Sorry, I can't follow you. No, 66. No, no, 65 was very... Για την 65 ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Πιστέψτε με. 66, το πρώτο τμήμα απορρίπτεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 και 68, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69, υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 78. Άρχεται. 78. The check is over. Πέρας. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές 83 Ο κύριος Βάλλη ε, επέμενε να γίνει ξεχωριστά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ Ο Μπάρτ ήθελε να ψηφιστεί ξεχωριστά. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε στην 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 102. Πέρας, απορρίπτεται. 103, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 105, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 108, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 108, παρακαλώ.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 24 α άλφα Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντα. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική σκέψη F υπέρ κατά. Α, όχι, όχι, όχι. Λέει η πρόεδρος. Λάθος έκανα. Εντάξει. Ψηφίζουμε. Τελική ψηφορία, ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφορία. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές. Και εγώ ψηφίζω υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Ήταν πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, πιστέψτε με. Και δεν είναι πρώτη φορά που οι υπάλληλοι της γραμματείας Κυριακή βράδυ συνέχιζαν τη δουλειά τους. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο στη μία. Ξέρετε όμως ότι ο συμβασμός είναι έθραυστος, γι' αυτό και θα παρακαλούσα, εν πάση περιπτώσει, ε, να στηρίξουμε τη γραμμή που ψηφίσαμε μόλις τώρα. Παρακαλώ. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Όλαφ, παρακαλώ ας αποχωρήσουν όσο, γίνεται πιο ήσυχα. Liebe Kollegin, liebe, ja, Συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε σας παρακαλώ. Όσο περισσότερο χρόνο σπαταλήσουμε τώρα, τόσο πιο αργά θα πάει η συνεδρίασή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μέρη σε διάταξη, ακρόαση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΛΑΦ 40 λεπτά έχουμε προβλέψει για κάθε υποψήφιο. Θα τους ακούσουμε αλφαβητικά και να υπενθυμίσω ότι μετά την ακρόαση θα γίνει μια, ένα μικρό διάλειμμα διαβούλευσης για τις πολιτικές ομάδες προκειμένου να γίνει αμέσως μετά απευθείας η ψηφοφορία. Καλύτερα τώρα παρά την Πέμπτη. Νομίζω ότι έτσι θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες. Ξεκινάμε με τον πρώτο υποψήφιο, τον κύριο Ήτελε τον οποίο και θα τον καλωσορίσουμε τώρα. Κάποιος ας τον καλέσει σας παρακαλώ. Πέντε λεπτά λοιπόν θα του δώσουμε για να μας συστηθεί και μετά θα ε, ακολουθήσει γύρω ομιλητών με βάση το σύστημα DONT. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ιτελα. Ah. Madam Chair, honourable members. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ο Όλαβ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν μιλούμε για αξιοπιστία και για εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Υπάρχουν Sorry. Is it okay? yes, it's okay. Sorry. Okay. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που μας απασχολούν. Εμπιστοσύνη, συνεργασία και χορήγηση κινήτρων. Και αυτά αλληλοσυνδέονται στενά. Σύμφωνα με την ε, πλέον πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλο μέρο των ε, Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Και ο Όλαφ ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο Όλαφ πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ε, εμπλεκομένων μερών και αυτό επιτυχάνεται μέσω καλύτερης και στενότερης συνεργασίας μαζί τους. Και όταν, λέω, όταν αναφέρομαι σε εμπλεκόμενους φορείς, εννοώ εσάς, την Επιτροπή Κοντ, τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και θέλω να πω εδώ και τώρα ότι το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες προκειμένου να μπορεί να εκτελεί τα, καθήκοντα, τα καθήκοντά του. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ πριν από 15 χρόνια περίπου ε, συμμετείχα στην, ε, στην, ε, στην ομάδα εργασίας δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων του Συμβουλίου και τότε ήδη είχαν ξεκινήσει συζητήσει. Εγώ ήμουν υπέρ τη δημιουργία και της θέσπισης αυτή τη ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 15 χρόνια μετά, επιτέλους έχουν ληφθεί τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει πλέον χώρο για αποτυχία. Από την αρχή λοιπόν, όλα και η ΕΠΟ χρειάζονται στενή συνεργασία και πρέπει να είναι σαφές ποιος κάνει τι, ποιος αποφασίζει τι, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις ή και ελλείψεις στο έργο των δύο οργάνων. Το έργο τους θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και να μεγιστοποιεί τις συνέργειες. Ένα από τα καλύτερα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μεταξύ των διευθυντών. Το νομικό πλαίσιο χρειάζεται αποσαφήνιση και εναρμόνιση. Για παράδειγμα, οι έρευνες για σημαντικά πρόσωπα, οι διαδικασίες και το παραδεκτό των ε, εκθέσεων του Όλαφ στα Εθνικά Συμβούλια. Πρέπει να τονίσω ότι ο Όλαφ θα παραμείνει ανεξάρτητος φορέας κεντρικής σημασίας. Με δύο λόγια, το όραμά μου για τον Όλαφ είναι να καταστεί ένα αμερόληπτο, διαφανές, σταθερό ηθικό, αποτελεσματικό, επαγγελματικό, ισορροπημένο και ελκυστικό θεσμικό όργανο. Όλες αυτές οι αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις και στο προσωπικό βεβαίως. Και το προσωπικό του Όλαφ είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. Είναι καθήκον μας να τους ακούσουμε, να τους, να τους ε, δώσουμε περισσότερες ε, ευκαιρίες κατάρτισης και επανεκπαίδευσης και να τους δοθούν ευκαιρίες ε, προαγωγής. Δεν χρειάζεται επανάσταση κυρία Πρόεδρε, πιστεύω όμως ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτιώσεων. Και τώρα να σας αναφέρω την εμπειρία που έχω. Από το 1984 στο 1988 ήμουν επικεφαλής εισαγγελίας ε, σε τρεις ε, περιφέρειες. Στη συνέχεια μεταπίδησα και έγινα δικηγόρος. Για ένα χρόνο. Στη συνέχεια εξελέγην στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο όπου προείδρευσα και σημαντικών επιτροπών. Στη συνέχεια έγινα Υπουργός Εσωτερικών και αναπληρωτής Πρωθυπουργός ιδιότητα με την οποία συμμετείχα και στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια εξελέγην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήμουν μέλο των Επιτροπών Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού και τα τελευταία χρόνια ε, θύτευσα στο Ελληνικό Συνέδριο. Ω άτομο είμαι πολύ επικοινωνιακό, ισορροπημένο και προσγειωμένο και δεν έχω καθόλου ε, συγκρούσει συμφερόντου από αυτή, την θέση μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ λέει η Πέτρη Σάβαμα, ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες. Έχουμε συμφωνήσει δύο λεπτά. Μία, ένα λεπτό ε, ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Ήταλα γιατί βρίσκεστε εδώ στην ακρόασή μας. Έχω δύο ερωτήσεις προς εσάς. Η πρώτη αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ρόλος και συνδεσιμότητα Όλαφ και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Όλαφ ε, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ε, που συλλέγει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και εσείς βλέπετε ότι χρειάζεται ίσως κάποια ανάγκη σε αυτή την επικοινωνία. Τώρα, ως προς τη διαφάνεια, Πώς βλέπετε τη διαφάνεια του Όλαφ, τι μπορεί να γίνει και πώς έχουν τα δικαιώματα αυτών που τελούν υπό έρευνα, που είναι ερευνόμενοι. Θα αλλάζατε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας ως προς το ελεγκτικό συνέδριο με ανησυχούσε αυτή η συνεργασία με τον Όλαφ, μεταξύ Όλαφ και ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί υπάρχει μηδενική σχεδόν συνεργασία. και έχουμε 500 τουλάχιστον ε, ελεγκτές in δεν υπάρχει ούτε κοινή εκπαίδευση, ούτε κοινέ συνεδριάσεις, ούτε ανταλλαγή προσωπικού. Δηλαδή, έχει σημασία να έχουμε μια επαφή με τους ελεγκτές οι οποίοι εργάζονται επί τόπου. Έχουν αυτή την εκπαίδευση να αναγνωρίσουν την απάτη. Αν λοιπόν συνεργαστούμε θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα είναι πολύ καλύτερη η συνεργασία. Τώρα θα έχουμε λιγότερους σπόρους από όσο γνωρίζουμε, γι' αυτό η συνεργασία είναι στοιχείο κλειδί για να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, μια δυναμική πορεία η οποία θα πρέπει και να αλλάξει. Ως προς τη διαφάνεια, σας είπα ότι μία από τις βασικές μου αξίες είναι αυτή στη Φιλανδία. Όταν συμμετείχα στην κυβέρνηση ε, επιδίωκα τη διαφάνεια διότι τα χρήματα του φορολογούμενου είναι πολύτιμα. Θα ήθελα να βελτιστοποιήσω την ε, διαφάνεια από πλευράς Όλαφ και μέσα στα πλαίσια της ε, ε, Εποπτικής Επιτροπής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος δράσης στο μέλλον. Ίσως υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει να είναι πραγματικά εξαιρέσεις. Και αυτό δεν αφορά τις έρευνες τη στιγμή που διεξάγονται. Η κυρία Αγιάλα, για ένα λεπτό. Σας ε, καλωσορίζω κυρία Ήταλα. Χαίρομαι γιατί πάντα συνεργαζόμασταν πολύ καλά στο παρελθόν, διότι στα πλαίσια του ελεγκτικού συνεδρίου είχαμε πολύ καλή συνεργασία και τώρα χαίρομαι γιατί είσαστε υποψήφιος να ε, μεταστραφείτε και να συμμετέχετε σε ένα πλαίσιο από το οποίο ξεκινήσατε, μέσα στα πλαίσια δηλαδή των ε, ελέγχων. Τι θα γίνει μέσα στα πλαίσια του υποπτικού μηχανισμού της Όλαφ, πέρα δηλαδή από το θέμα του προσωπικού, θα ήθελα να ρωτήσω πώς έχει αυτή η σχέση με την Επιτροπή Εποπτείας από το ελεγκτικό συνέδριο κρίνεται όλα πολύ περισσότερο από ότι προωθείται μία συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ερευνόμενους. Θα ήθελα να μας πείτε μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαίου Ισαγγελέα πώς θα εξελιχθεί αυτός ο ρόλος μέσα στα πλαίσια του κυρωτικού μηχανισμού και πώς θα μπορέσετε να δράσετε ως αστυνομική αρχή έτσι ώστε ο Όλαφ να μπορέσει να δράσει υπό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εσείς βλέπετε ένα μέλλον σε αυτή τη συνεργασία. Θεωρείτε ότι στο μέλλον ε, η Όλαφ θα μπορέσει να πείσει όλες τις χώρες προς αυτή την κατεύθυνση ότι δηλαδή ο Ευρωπαίος εισαγγελέα θα μπορούσε να προβάλλει μια συνεργασία και με την Όλαφ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, ως προς τον, ε, την εποπτική αρχή και την Εποπτική Επιτροπή θα ήθελα να ενισχύσω το ρόλο της Πρωτίστως, όπως προείπα, θα πρέπει να δώσουμε όλες τις πληροφορίες, εκτός από αυτές που αφορούν την ε, περίοδο της έρευνας, για να δούμε πώς θα μπορέσουν να δράσουν και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Εγώ προέρχομαι από ε, έναν εποπτικό μηχανισμό και αρχή. Άρα καταλαβαίνω ότι μόνο με, την, με τις επικρίσεις μπορεί κανείς να βελτιωθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε στενή συνεργασία. Δεν πρόκειται μόνο για εποπτεία. Μπορούν να ασκήσουν και ε, συμβουλευτικό ρόλο υπομορφή ε, δεοντολογικών αρχών. Εάν εκλεγώ θα ζητήσω τη γνωμοδότησή τους. Τσαρνέτσκι, για ένα λεπτό. Δεν ε, θέλετε το λόγο, σας είχα στον κατάλογο κανένας από το ECR. Λοιπόν, ε, φιλελεύθεροι. Σας ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Ιταλά. Η μία ε, ερώτηση απαντήθηκε γιατί θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, Εποπτική Επιτροπή ε, γιατί η Επιτροπή λυπάται για το γεγονός ότι η Όλαφ δεν επιτρέπει πρόσβαση στα στοιχεία της από την ε, ε, Επιτροπή Εποπτείας. Θα μπορέσετε να προωθήσετε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία ή θα υπάρχουν ε, περιορισμοί. Και το δεύτερο ερώτημα, έχετε μία μακρά σταδιοδρομία και στη Φιλανδία και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ποιες είναι ε, οι δύο βασικότερες ε, πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλάβατε στην ε, πολιτική σας δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια των δύο αυτών ρόλων. Σας ευχαριστώ πολύ για να είμαστε συγκεκριμένοι. Φυσικά η παροχή πληροφοριών είναι ύψης της σημασίας εγώ θα παράσχω όλες τις πληροφορίες μέσα στα πλαίσια του, των ε, νομικών δεσμεύσεων, αλλά όχι εκεί που διενεργείται έρευνα. Όταν κλείσει η υπόθεση, τότε θα μπορέσει η Εποπτική Επιτροπή να έχει όλες τις πληροφορίες, ε, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε εγγύηση ε, αυτονομίας και ανεξαρτησίας της Όλαφ, ιδιαίτερα όταν ανοίγουν υποθέσεις και όταν λήγουν ή αποσύρονται υποθέσεις. Γιατί διαφορετικά, εάν δεν παρασχέται όλες, όλες τις πληροφορίες, τότε κανείς πέσει με στατιστικά στοιχεία όταν δεν διαθέτει πληροφορίες θα πρέπει να βασιστεί σε στατιστικές, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Θα ήθελα να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την ε, Εποπτική Επιτροπή. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συμμετείχα και εγώ. Ήμουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά υπάρχουν ε, συμφωνίες και διαφωνίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Στάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισέλθουμε περαιτέρω Καταρχά να σας καλωσορίσω, γνωριζόμαστε και από παλιά. Θα ήθελα να εξετάσουμε τη δύσκολη σχέση που ε, παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια μεταξύ του προηγούμενου Γενικού Διευθυντή του Όλαφ και της Εποπτικής ε, Επιτροπής. Είπατε μόλις, απαντώντας στα ερωτήματα της Μαρτίνα, ότι θα είστε πολύ ανοιχτός ως προς την Επιτροπή. Όμως, εάν διοριστείτε ως νέος Γενικός Διευθυντής, θα συνεργαστείτε πλήρως, είπατε, με την Επαπτική Επιτροπή και θα διασφαλίσετε τους ώστε να υπάρχει γενική και απόλυτη διαφάνεια, φυσικά για αυτούς τους φακέλους που έχουν κλείσει, ε, για να φανεί αν όντω έχουν εξεταστεί σωστά από την Όλαφ. Επομένως, μας λέτε ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και θα είστε απόλυτα ανοιχτός απέναντί μας. Μάλιστα, είπα και προηγουμένως ότι η διαφάνεια είναι μία από τις ε, βασικές αξίες. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που μου επιτρέπεται από τον νόμο να σας δώσω. Όλες οι πληροφορίες, λοιπόν, που δεν ε, σχετίζονται με ε, έρευνες που ακόμα δεν έχουν κλείσει. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ. Βέβαια δεν είναι η δική μου απόφαση, αλλά θέλω να ενισχύσω και το ρόλο της Επιτροπής αυτής για να εργαστεί και ως δεοντολογική επιτροπή. Δηλαδή όχι μόνο να παίρνουν τις ε, πληροφορίες και να ε, γνωμοδοτούν ε, σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε δεοντολογικό Υπάρχει αυτή η πρόταση του ελεγκτή για τον Όλαφ εγώ δεν είμαι υπέρ. Γιατί να δημιουργήσουμε νέα επίπεδα, νέες δομές. Ήδη έχουμε μια πολύ καλή και επαγγελματική ε, εποπτική επιτροπή. Σε αυτή λοιπόν θα πρέπει να βασιστούμε και η Όλαφ ε, υποχρεούται να δώσει όλες τις πληροφορίες ε, που πρέπει. Ο συνάδελφος Δεγιόμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά αυτή την ελεγκτική ιδιότητα και, την, και η Εποπτική Επιτροπή βέβαια μπορεί να κάνει πολύ καλό έργο αν λάβει και περισσότερες αρμοδιότητες σε αυτό το πεδίο. Πολλά κράτη-μέλη λένε ότι δεν χρησιμοποιούν τους ελεγκτές της Όλοφ γιατί είναι ασαφείς οι διαδικαστικοί κανόνες ή δεν συνάδουν με την ε, νομοθεσία του κράτους μέλους. Όμως, τι θα κάνετε για να μεριμνήσετε για την προάσπιση της ποιότητας και των αξιών που υπερασπίζεται ε, ο Όλαφ. Εσείς δεν έχετε εμπειρία στον τομέα της έρευνας, οπότε τι ρόλο θα δραματίσετε σε αυτό το πλαίσιο. Μετά, για την ε, διαχειριστική ιδιότητα. Από πλευράς λοιπόν ε, διαχείρισης, τι είδους εμπειρία έχετε. Uh, Αν κατάλαβα καλά. Με ξαναρωτήσατε για την ε, Εποπτική Επιτροπή και πώς αυτό συνάδει με τις διαδικασίες και τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη Πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, αλλαγές ε, στο κανονιστικό πλαίσιο για να δουλέψει αυτό το σύστημα καλά. Οι ενδιαφερόμενοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ε, πρόσβαση στους φακέλους του Όλαφ. Βλέπουμε ότι οι διοικητικέ έρευνες δεν είναι τόσο ισχυρές. Εγώ διαφωνώ. Σε σχέση δηλαδή με, με την ποινική εξέταση. Γιατί πρώτα έχουμε τη διοικητική έρευνα και μετά, ίσως από δύο χρόνια, να περάσουμε ε, στο ποινικό σκέλος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να περιμένω ενδιαφερόμενος. Μία από τις ε, βασικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι δικαιούνται μια δίκαιη δίκη. Πώς όμως μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για αυτή την ε, δικαιή δίκη αν δεν γνωρίζει τις ε, λεπτομέρειες της υπόθεσης. Και η δίκαιη δίκη δεν ξεκινάει κατά την έναρξη της δίκης, αλλά πολύ πριν κατά την προετοιμασία της δίκης. Ελπίζω λοιπόν ε, να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο. Εντάξει, τώρα με την Ευρωπαϊκή Συγγελία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αλλά πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και αποσαφήνιση του κανονισμού. Οι ε, ελοχεύουν κίνδυνοι. Ο συνάδελφος Βάλλη. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για τον υποψήφιο. Πρώτον, πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε τις σχέσεις ε, του Όλαφ και των κρατών μελών. Υπάρχουν μία σειρά συστάσεις που δεν γίνονται σεβαστές. Θα ήθελα να δω ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις για να καταλήξετε σε κάποιον συμβιβασμό, παρότι καταλαβαίνω ότι από πολιτική άποψη αυτό δεν είναι εύκολο. Και ποιος θα είναι ο ρόλος του Όλαφ ε, ως προς τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. πώς θα γίνονται οι έρευνες προς αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων, για παράδειγμα. Εξετάζοντας το βιογραφικό σας, είδα ότι έχετε και μακρά πολιτική σταδιοδρομία. Θα ήθελα λοιπόν να δω τι ε, είδους εχέγγυα μπορείτε να δώσετε για την αμεροληψία σας στη θέση του ε, Γενικού Διευθυντή, καθώς έχετε και πολιτική ιστορία. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω. Πρώτα για τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντικά τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι ζωτική σημασία λοιπόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτά τα λεγόμενα αύκος σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το παραδεκτό των ε, εκθέσεων του Όλαφ είναι σημαντικό θέμα. Απαιτείται λοιπόν ε, ενισχυμένη συνεργασία. Όπως είπα, το πιο σημαντικό μέσο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Το πώς θα γίνει, ε, καλό είναι να ξεκινήσουμε σε επίπεδο διευθυντή και ίσως στη συνέχεια να περάσουμε στους εξωματικούς συνδέσμους. και δεν έχουμε περιθώριο βεβαίως να αποτύχουμε εδώ. Απαιτείται πραγματικά στενή συνεργασία και απόλυτη διαφάνεια. Γιατί μπορούμε εδώ να αρχίσουμε τα ευχολόγια, όμως ε, στην πράξη θα πρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Ζακ. Ε, ε, Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ε, θέσω το εξής ερώτημα. Πρόσφατα μάθαμε κάτι το οποίο μας λείπησε ιδιαίτερο, ε, ότι απεβίωσε ο κύριος Τωτορίνα, που ήταν ηθήνων ε, νους της μαφίας της Καλαβρέζικης. Ε, είδαμε μια σειρά ρεπορτάζ και πραγματικά έμεινα άναυδος όταν είδα ένα ρεπορτάζ στην γαλλική τηλεόραση. Μπορώ να σας δώσω και τις λεπτομέρειες. Ότι κάποια στιγμή έχουμε ένα νέο 35 ετών που... κανονικά θα συνέχιζε ε, την και θα γινόταν επικεφαλής αλλά μετά ε, μετανόησε και άλλαξε ε, ρότα και αναφέρθηκε ότι η μαφία στην ε, Καλάμπρια έχει υπεξαιρέσει ποσά στις τάξεις των δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρείται ότι τέτοιου είδους υπεξαιρέσεις θα αποτελέσουν προτεραιότητα για τον οργανισμό σας. Uh, Μάλιστα, αν ε, εκλεγώ, η παριθμόν ένα προτεραιότητά μου θα είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, που βέβαια άπτεται αυτού που αναφέρατε. Γιατί συνεχώς αλλάζουν οι συνθήκες ε, και οι εγκληματίες συνεχώς ε, βελτιώνονται και εξυγχρονίζονται. Απαιτείται λοιπόν πολύ καλή συνεργασία με όλου του εμπλεκόμενου φορεί, αλλά και χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα. Οι εθνικές ε, αρχές βλέπω ότι ε, χρησιμοποιούν πλέον νέε μεθόδους ε, επεξεργασίας δεδομένων. Δεν είμαι ειδικό, αλλά το είδα με τα μάτια μου και από ό,τι βλέπω, εάν κανείς έχει ένα σύνολο δεδομένων, από το δικαστήριο του Eurojust, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνει κανείς όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις παρατυπίες και την απάτη. Και αν δείτε την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, ε, είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο. Και αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ο συνάδελφος Λαφράγκα. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι που είναι μεταξύ μας ο πρώην συνάδελφος Ήταλα. Έγινε λόγος για τις ε, διαχειριστικές του ικανότητες. Ξέρουμε ότι ήσασταν υπουργός, διατελέσατε υπουργός και φυσικά εκπροσωπήσατε τη χώρα σας στο Συμβούλιο Υπουργών Εργαστήκατε στο ελεγκτικό συνέδριο και συμμετείχατε ως Ευρωβουλευτής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε λόγος για τα ε, δικαιώματα παροχής πληροφοριών για τους ερευνόμενους και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να χορηγούνται οι πληροφορίες κατά τη ε, διενέργεια της έρευνας αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι η ενδεχόμενη ε, συνεργασία με την Εποπτική Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο στο μέλημά σας. Ευχαριστώ. Ως μέλος της Επιτροπής ΚΟΝΤ, πρώην μέλος, γνωρίζω πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία και ως ε, εμπλεκόμενος και συνδεδεμένος φορές με, την, τον Όλαφ, η Κοντ, είναι ο μόνος εκπρόσωπος των πολιτών. Ο μόνος άμεσα αιρετός εκπρόσωπος των πολιτών. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική η Επιτροπή σας. Εγώ σκοπεύω να έρχομαι, να σας επισκέπτομαι ε, όσο συχνά επιθυμείτε εσείς και να οικοδομήσουμε και προσωπικές ε, σχέσεις γιατί η εμπιστοσύνη ε, στον Όλαφ είναι ύψης της σημασίας είναι πρώτη προτεραιότητα η συνεργασία αυτή και θέλω να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη όποιο και αν είναι το τίμημα. Γιατί μέσω ημών με ύψιλον μπορούμε να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών στον Όλαφ. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ήτελε, Είστε ένας από τους τέσσερις υποψήφιους. Έχετε πραγματικά εντυπωσιακό βιογραφικό. Έχετε εργαστεί στην Επιτροπή Προπολογισμών, σε άλλους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς και θα θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει τα ζητήματα ε, που σχετίζονται με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Ε, δυστυχώς, τέτοιου είδους συστήματα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως ο Όλαφ δεν έχει πρόσβαση στα συστήματα αυτά. Συστήματα που σχετίζονται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ιδίω όταν σκεφτόμαστε την ε, ε, καταπολέμηση των ριζικών αιτίων και όχι μόνο των συνεπειών ορισμένων προβλημάτων. Δεύτερο ερώτημα. Ο Όλαφ είναι οργανισμός που δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της Κομισιόν. Είστε ε, ευχαριστημένος με την έως τώρα συνεργασία του Όλαφ με την Κομισιόν και τι σκοπεύετε να ε, κάνετε στο μέλλον σε σχέση με αυτό το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό αυτή η κοινή βάση δεδομένων είναι απαραίτητο να υπάρξει. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ακριβώ για να δημιουργηθεί αυτή η κοινή βάση δεδομένων με κοινά δεδομένα, κάτι που θα αποτελέσει το καλύτερο δυνατό εργαλείο για την καταπολέμηση παρατυπιών. Φυσικά, χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεται να γίνουν συζητήσει με όλα τα κράτη-μέλη λόγω του ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα, διάφορες δομές, διάφορα επίπεδα ε, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Για τη συνεργασία με την Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως, ο Όλαφ αποτελεί τμήμα της Κομισιόν, αλλά διοικητικά ε, χρειάζεται καλή συνεργασία προφανώς. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι όταν διεξάγεται έρευνα δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία για την αμεροληψία του οργανισμού αυτού. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι δηλαδή ο Όλαφ ε, ενεργεί ε, αμερόληπτα όταν διεξάγει έρευνες. Ο Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ιτέλε για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήματα να σας θέσω. Πρώτον, Τι σκοπεύετε να κάνετε σχέση με, με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων του Όλαφ. Γνωρίζουμε ότι ο Όλαφ ε, προσελκύει παραδοσιακά τους καλύτερους ε, στον τομέα της ε, καταπολέμησης της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς θέλετε εσείς να σχιστεί αυτή η παράδοση. Δεύτερο, γιατί εμείς οι ευρωβουλευτές δεν λαμβάνουμε τις εκθέσεις του Όλαφ ή έστω κάποιες περιλήψεις αυτών των εκθέσεων. Δεν μας τις παρουσιάζεται. γιατί ο Όλαφ ε, έχει μείνει τόσο πίσω ως προς την επικοινωνία του με το κοινό. Θέλετε να κάνετε κάτι προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως είπα, το προσωπικό του Όλαφ είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Είναι σημαντικό να νιώσει κάθε εργαζόμενος του Όλαφ ότι αποτελεί μέρος της ομάδας. Αυτό κάνω εγώ πάντοτε στη ζωή μου. Είμαι ε, άνθρωπος που μου αρέσει να εργάζομαι σε ομάδες και θέλω κάθε υπάλληλο του Όλαφ να έχει την ίδια αίσθηση. Ο διευθυντής έχει ως καθήκον να καταδείξει την κατεύθυνση του οργανισμού αλλά ταυτόχρονα να δώσει κίνητρα ε, και να ενθαρρύνει, να παροτρύνει τους εργαζόμενους του προκειμένου να κινηθούν και εκείνοι σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και μίλησα για περαιτέρω ε, δυνατότητες κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και προαγωγής των υπαλλήλων. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες στον Όλαφ ότι 45 άνθρωποι θα μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη συνέχεια τι όμως τι θα γίνει. Θα προσληφθούν 20 νέοι, 40 νέοι, θα μείνουν και νέες αυτές οι θέσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να δοθεί μια υπόσχεση από εδώ ότι τελείωσε. 45 άνθρωποι θα μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελειώσαμε. Ότι δεν θα γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε χρόνο. Ευχαριστώ ο κύριος Πυρίντσκι. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι κύριε Ήτελε. Εδώ. Στα αριστερά σας. Ένα λίγο ευρύτερο θέμα θέλω να θίξω εγώ. Στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας και της θητείας της Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην δημοσιευθεί η Γενική Έκθεση για τη Διαφορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντιθέτως να ε, αντιμετωπίσει ζητήματα διαφοράς αναχώρο χώρα, ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είπατε και εσείς ο ίδιος ότι οι περισσότερες παρατυπίες και φαινόμενα ε, διαφοράς είναι διασυνοριακές το ερώτημά μου λοιπόν που με έχει απασχολήσει προσωπικά ε, επί μακρόν είναι ότι υπάρχει κάποια ε, ε, υπόθεση εργασίας ότι κάποιες χώρες είναι πιο διεφθαρμένες από άλλες. Ιδίως αναφέρομαι σε χώρες όπως η Βουλγαρία ή εν γέννη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα ε, συστήματα, από αυτά, από αυτά τα κυκλώματα ε, έχουν την αφετηρία τους και την πηγή τους ε, σε, σε, σε παλαιά κράτη-μέλη. Εσείς πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε την αμεροληψία σας και να, για να μπορείτε να εξετάζετε το κάθε περιστατικό, την κάθε υπόθεση στο πλαίσιό της, χωρίς να θεωρείτε δεδομένο ότι ε, κάποιες χώρες ε, πλήττονται περισσότερο από άλλες από το πρόβλημα της διαφθοράς. Απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό όποιος κι αν ε, εκλεγεί διευθυντής, γενικός διευθυντής του Όλαφ, να μην θεωρεί να μην έχει τέτοιες προκαταλήψεις απέναντι σε συγκεκριμένες χώρες. Πρέπει να κάνει επαγγελματικά τη δουλειά του, όποτε λοιπόν εμφανίζονται υποθέσεις, να συλλέγει στοιχεία προκειμένου να ξεκινά η έρευνα. Δεν μπορεί να σκέφτεται ένας γενικός διευθυντής με αυτόν τον τρόπο ότι μια χώρα είναι χειρότερη από την άλλη. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε θα χάσεις και τον προσανατολισμό σου αν ε, κάνεις κάτι τέτοιο. Ε, αν θεωρείς δηλαδή ότι κάποιες χώρες είναι χειρότερες από άλλες. Πρέπει να εξετάζεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και όχι να βάζεις ε, τα κράτη-μέλη ε, σε κάποια ιεραρχία, ε, σε κάποια κουτάκια ανάλογα με το πόσο διεφθαρμένα ή όχι θεωρεί, ότι, θεωρείς ότι είναι. Ο κύριος Νόβακο. Ευχαριστώ. Κύριε Ιταλά, έχοντας κατά νου την εμπειρία, την εμπειρία σας ως Υπουργού Εσωτερικών και Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, Πιστεύετε ότι οι αρμοδιότητες του ΟΛΑΦ πρέπει να διευρυνθούν όσον αφορά τις λειτουργίες του οργανισμού αυτού, διότι στις μέρες μας ο Όλαφ ε, μπορεί να εντοπίσει ε, παρατυπίες σε σχέση με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ταυτόχρονα όμως εξαρτάται από τις εθνικές αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν την έρευνα και να εκπληρώσουν τη διαδικασία, να προσφύγουν στα δικαστήρια κτλ. κτλ. Δεύτερο ερώτημα. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαίου Σαγγελέα και πώς μπορεί να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεργαστεί με τον Όλαφ. Ακριβώς γιατί τα ζητήματα που θα αποσχολούν και, τους, και τα δύο όργανα θα είναι ευρωπαϊκά. Αντιστοίχω λοιπόν ευρωπαϊκές θα πρέπει να είναι και οι λύσεις. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η συνεργασία των δύο οργάνων. Πρώτον, όσον αφορά την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του Όλαφ. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια τέτοια διεύρυνση. Και θα σας πω και συγκεκριμένα. Υπάρχουν δύο ε, που είναι πολύ κρίσιμης σημασίας. Πρώτον, πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις ε, ροές κεφαλαίων. Όταν διεξάγει κανείς μια έρευνα ε, με αντικείμενο χρηματοοικονομικά εγκλήματα και δεν μπορείς να έχεις καν πρόσβαση ε, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πώς μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ πραγματικά εξεπλάγει όταν έμαθα ότι ο Όλαφ δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει ε, και να απευθυνθεί στι τράπεζες για να λάβει πληροφορίε. Αυτό και ε, βεβαίως το παραδεκτό των εκθέσεων του Όλαφ στα εθνικά δικαστήρια. Γιατί μπορεί ο Όλαφ με βάση το σημερινό πλαίσιο να ε, δουλέψει δύο χρόνια πάνω σε μια υπόθεση και στη συνέχεια όταν τελικά καταλήξει η υπόθεση στα εθνικά δικαστήρια η έρευνα πρέπει να ξανά γίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αυτά τα δύο δηλαδή. Πρόσβαση ε, τραπεζικούς λογαριασμούς ε, και αυτό συνδέεται και με το ΦΠΑ όπου ε, πρέπει πραγματικά ο Όλαφ να αποκτήσει τη δυνατότητα, τη νομική, να, και, να ερευνά και τέτοιου είδους υποθέσεις. Ο κύριος Κον, ευχαριστώ. Ακριβώς ε, το ίδιο θέμα θέλω να θέσω κι εγώ. Ιδίως ε, στον φόρο προσθέμενης αξίας υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και του Όλαφ σε περιπτώσεις απάτης. Εσείς πώς θα προσπαθήσετε σε αυτές τις υποθέσεις να αποφύγετε αυτόν τον ανταγωνισμό και να επιτύχετε ε, την επίτευξη κοινών στόχων. Να καταπολεμηθεί δηλαδή η απάτη και η διαφθορά χωρίς ωστόσο να ανταγωνίζεται όλα τις εθνικές αρχές. Ναι, είπα ότι αυτό θα πρέπει να διασαφινιστεί στον κανονισμό προς τον ε, ΦΠΑ αφορά το θέμα της προστασίας οικονομικών συμφερόντων. Πρόκειται για την οδηγία PIF και νομίζω ότι ο ΦΠΑ υπάρχει στον κανονισμό, αλλά στην περίπτωση του Όλαφ, τι θα γίνει εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, ζητήσει από τον Όλαφ να συνδράβει σε ορισμένες έρευνες. Θα πει ο Όλαφ ότι αυτό δεν εντάσσεται στην εντολή μας. Νομίζω ότι αυτό χρήζει διασαφήνισης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη διότι παρατήρησα ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν αυτή τη ε, ε, διασαφήνιση στον κανονισμό του Όλαφ. Ε, χρειάζονται διαπραγματεύσεις λοιπόν διότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε επίπεδο Συμβουλίου γιατί ίσως να μην συμφωνήσει το Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του ΕΛΚ. Θέλω να ε, επανέλθω σε ένα ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ντεγιόμ και αφορά την εμπειρία, τη διαχειριστική. Ε, τι είδου εμπειρία έχετε σε διευθυντικές θέσεις και το δεύτερο αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα των οίκων συμψηφισμού. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, στα πλαίσια της ε, διαχείρισης του ΟΛΑΦ, είδα αυτή την διάρθρωση του ΟΛΑΦ και είδα ότι υπάρχει μια τέτοια ε, διάρθρωση ε, προτεραιοτήτων μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στο ελεγκτικό συνέδριο. Είδαμε ότι ε, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος εργασίας αυτός, δεν είναι ευέλικτος. Γι' αυτό επειδή δεν συμμετείχα στον Όλαφ, δεν ξέρω πώς ε, λειτουργεί αυτό το πλαίσιο, αλλά αν, θέλει κανείς να τα ελέγξει αυτά γρήγορα και να τα εντάξει σε μία πορεία, τότε θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω αν ε, προϋπάρχει αυτή η διάρθρωση συνεργασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι πιο αποτελεσματικός ο Όλαφ για να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. γιατί θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα σε μια τέτοια περίπτωση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έχουμε πείρα σε αυτό το τομέα. Ως προς το, τα γραφεία συμψηφισμού έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που έχει ε, σημασία είναι ε, να υπάρχει συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βεβαίως ε, δεν είναι εμπλεκόμενος φορέας η Κομισιόν γιατί όλα Όλαφ εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, έληξε λοιπόν η ακρόαση του πρώτου υποψηφίου. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα, ο, συνάδελφος, μάλλον, ο συνάδελφος Κάλφιν, ο υποψήφιος, ο κύριος Κάλφιν είναι παρόν. Ja, wir machen weiter mit einem uns ebenfalls sehr gut bekannten früheren Kollegen, Kollegen Evailo Kalfin. Ε, γνωρίζετε πολύ ε, καλά τον πρώην συνάδελφο, τον ε, κύριο Κάλφιν. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, κυρίε και κύριοι, αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να διαδραματίσει ενεργό ρόλο όχι μόνο στην επιλογή ε, του επόμενου Γενικού Διευθυντή, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του μέλλοντο αυτού του οργανισμού με σκοπό, που έχει ω σκοπό την προστασία των οικονομικών σφαιρόντων τη Ένωση και των πολιτών, καθώ και την ακαιρεότητα των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Έχω την τιμή να παρουσιάσω τις απόψεις μου ε, εδώ και την υποψηφιότητά μου μαζί με τρεις ακόμα αξιότιμους συναδέλφους. Είναι πραγματικό προνόμιο για μένα. Όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι βασικές αξίες ε, του Όλαφ, ε, ποια είναι η εντολή του οργανισμού αυτού. Πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες και να ε, συνεργάζεται με μια σειρά φορέων. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα εύρωστο σύστημα για την καταπολέμηση τη απάτη, παρά τα θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Ο Όλαφ όμω δεν κατάφερε ε, να διατηρήσει απόλυτα διαφανεί σχέσει με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά μια σειρά έρευνε. Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του ε, επόμενου Γενικού Διευθυντή είναι η αποκατάσταση του διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ε, μπορεί όλα Όλαφ να είναι ισχυρός, αποτελεσματικός, αλλά και διαφανής ε, φορέας για την τήρηση των αξιών που θέλουμε, για την προάσπιση των συμφερόντων ε, στα δημόσια οικονομικά. Η Εποπτική Επιτροπή θα είναι πολύ σημαντική. γιατί εμείς κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων ε, μπορώ να επισέλθω ε, σε προς λεπτομέρειες. Βασική προτεραιότητα για τη νέα ηγεσία θα είναι η θέσπιση ε, καλών σχέσεων εργασίας με τη νέα Ευρωπαϊκή Συγγελία που θα συσταθεί του χρόνου. Δεν υπάρχει ε, καμία αντιπαλότητα μεταξύ των δύο. Η σύσταση της εισαγγελία είναι πολύ σημαντικό βήμα ε, που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των φορολογουμένων ε, και μας επιτρέπει την σωστή καταπολέμηση της απάτης. Θα είναι αυτό η σιδηρά χείρα που θα φέρει όλες αυτές τις υποθέσεις απάτης ενώπιον της δικαιοσύνης. Απαιτείται ε, ισχυρή στήριξη από όλες τις πλευρές και από τον Όλεφ. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη για να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Συγγελία. Εν τω μεταξύ, Παράλληλα με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αγγελία και όλα μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι εσωτερικό φορέας που συνεργάζεται με όλα τα κρατημέλη και έχει πρώτης ε, τάξεως ε, ερευνητικό προσωπικό εξετάζει ζητήματα ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού αλλά και υποθέσεις σοβαρή ε, σοβαρής κατάχρησης εξουσίας Ευρωπαϊκού στους ευρωπαϊκούς Είναι λοιπόν ένα από του φορεί που καταπολεμά την απάτη και έχει μοναδικές αρμοδιότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την προστασία των σφαιρών των πολιτών πρέπει να προσδιορίσουμε πολύ συγκεκριμένα τις ε, αρμοδιότητες του Όλαφ και της ε, εισαγγελία, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Όλαφ θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να, διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα εξή τρία στοιχεία. Να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις ε, ερευνών μεταξύ των δύο φορέων. ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών, αμφίδρομη και να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια που τυχόν απομένουν. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, οπότε περιμένω τα ερωτήματά σας. Πέραν ε, της θέσπισης αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Όλαφ και της ε, Ευρωπαϊκής Συγγελίας, απαιτείται και μια πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την, μάλλον την ε, Εποπτική Επιτροπή. Στόχος μου θα είναι να ενισχύσω την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και να εισαγάγω νέες τεχνολογίες ε, στην εκτέλεση και τον έλεγχο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Όλο το σύστημα καταπολέμησης της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο κατόφλι μιας μεγάλης αλλαγής. Και νομίζω ότι η έρευνα δεν είναι το βασικό μέλημα αυτή τη στιγμή για τον Όλαφ, γιατί υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί ερευνητές. Το βασικό ζήτημα είναι ε, η σωστή εμπλοκή του Όλαφ ε, στο όλο σύστημα καταπολέμησης της απάτης και η ενεργός προβολή του, προκειμένου να καθησυχάσουμε και τους πολίτες ότι προασπίζονται ε, οι ευρωπαϊκοί φορείς ε, τα συμφέροντά τους. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό θεσμικό όργανο που θα δράσει ως πραγματικός εγγυητής των, δικαιωμάτων, των συμφερόντων των πολιτών. Είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να εκπληρώσω αυτά τα καθήκοντα. Στη σταδιοδρομία μου έπρεπε πάντα να ε, τηρώ στενά χρονικά περιθώρια, να διατηρώ την ακεραιότητά μου παρά τις ε, πολιτικές πιέσεις ε, και να κάνω το καλύτερο δυνατόν παρά την διάσταση των πολιτικών συμφερόντων. Γνωρίζω τα του προπολογισμού από πολλές διαφορετικές πλευρές και Έχω βαθιά γνώση του ενωσιακού προπολογισμού και η δημοσιονομική πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, κατανομή, αλλά και την αποτελεσματικότητα ε, των δημοσίων οικονομικών και την, την παροχή εχεγγύων προς ε, τον φορολογούμενο. Η εμπειρία μου, οι γνώσεις μου και το ιστορικό μου μου δίνουν την πεποίθηση ότι αν εκλεγώ θα είμαι ένας πολύ καλός γενικός διευθυντής του Όλαφ. Θα λαμβάνω υπόψη τα επιτεύγματα και ε, θα συνεχίζω με βάση τις νέες προκλήσεις. Δεν, δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις που κατήχα. Ε, κυρία Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, σας ευχαριστώ και πάλι για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το όραμά μου για τον Όλαφ και είμαι στη διάθεση για τυχόν ερωτήσεις. Ε, ήμουν και μέλος ε, της Επιτροπής Κόντ και γνωρίζω το υψηλό επίπεδο που σας χαρακτηρίζει. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Άβαμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλφιν για την παρουσία σας εδώ. Μπορεί να μην με, να με θυμάστε, εγώ όμως σίγουρα σας θυμάμαι από το παρελθόν. Πρώτον, είναι πολύ ενδιαφέρον ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ή μάλλον για να το θέσω καλύτερα, έχει ρόλο το ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά τις έρευνες. Ο Όλαφ αξιοποιεί μέχρι στιγμής τις πληροφορίες που διατηρεί το ελεγκτικό συνέδριο. Και είναι κάτι το οποίο σκοπεύετε να αλλάξετε με οποιοδήποτε τρόπο ως γενικό Διευθυντής. Δεύτερο ερώτημα για τη διαφάνεια. Πώς θα χειριστείτε το ζήτημα της διαφάνειας ως Γενικός Διευθυντής του Όλαφ και ποιος, ε, πώς πιστεύετε ότι ε, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ερευνόμενων στο πλαίσιο της διαφάνειας και της εκτέλεσης των καθηκόντων του Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάββαμα. Πρώτον, για τον ρόλο του ελληνικού συνεδρίου. Πρόκειται για δύο φορείς ε, του ίδιου μηχανισμού καταπολέμησης ε, της απάτης ε, όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση που έλαβε το ελεγκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο ορίζει και το πλαίσιο διασύνδεσης και συνεργασίας των δύο φορέων. Αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και ε, τον τρόπο χειρισμού πληροφοριών που έρχονται σε γνώση του ενός ή του άλλου και καθορίζει ε, τον τρόπο και τους όρους για την αποκάλυψη ε, συγκεκριμένων πληροφοριών. Θεωρώ ότι ο μηχανισμός αυτός είναι θετικός, αλλά θεωρώ ότι θα χρειαστεί να συζητήσουμε περισσότερο τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Όλαφ με συναδέλφους σας που ε, ισχυρίζονται κάποιες φορές ότι ο Όλαφ δραστηριοποιείται στα όρια της νομιμότητας ε, ιδίως όσον αφορά την εκ των προτέρων διερεύνηση υποθέσεων από την πλευρά του Όλαφ αλλά και τις διαδικαστικές κατευθυντήρες γραμμές που τηρούνται ή δεν τηρούνται ορισμένες φορές. Μιλώντα λοιπόν για το ρόλο και τη διάδραση μεταξύ του ελεγκτικού συνεδρίου και του Όλαφ υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ξεκοθαριστούν και νομίζω ότι η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, είναι θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και ε, ειδικέ εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου για τη δραστηριότητα του Όλαβ. Υπάρχουν και συγκεκριμένα νομικά ζητήματα που έχουν τεθεί και αναλυθεί αλλά ε, για τον Όλαφ συνολικά, αλλά και για το Εποπτικό Συμβούλιο και ε, νομίζω επίσης ότι πρέπει να αναπτυχθούν και κάποιες διαδικαστικές εγγυήσεις προκειμένου να ε, διαμορφωθεί ε, το πλαίσιο της συνεργασίας. Για τη διαφάνεια θα μου πείτε κάτι. Όχι, λέει η Πρόεδρος, επεμβαίνοντας Έχετε ήδη απαντήσει μαζί με την ερώτηση δύο λεπτά. Η κυρία Αγιάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο ε, Κάλφιν, ο οποίος ε, έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό και ως πρώην Υπουργός ε, και στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά σε όλες τις ε, δραστηριότητες και μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής ε, Ιδίων Πόρων όπου συμμετείχε και ο κύριος Μόντι. Όπως ξέρετε με την κυρία Γκρέσλε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διελκυστίνδας ως προς αυτό το θέμα ιδιαίτερα ως προς την απάτη για το ΦΠΑ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε αυτό το πλαίσιο εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης, ιδιαίτερα στις όμορες περιοχές. Πώς θεωρείτε ότι ένας γενικός διευθυντής του Όλαφ θα μπορούσε να ε, άρει αυτούς τους σκοτεινούς ε, διαδρόμους ε, ως προς τους, ε, τη διαχείριση των ιδίων πόρων. Με τα εθνικά κοινοβούλια επίσης υπάρχει συνεργασία, αλλά όταν μεταβαίνουν μέλη του Όλαφ σε κράτη-μέλη φαίνεται ότι εκτροχιαζόμαστε από το σωστό πλαίσιο εργασίας. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν παρακολούθηση αυτών των ε, φακέλων μέσα στα πλαίσια των Εθνικών Αρχών και του Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ε, αφορά και απάντηση στην προγενέστερη ερώτηση. Η διαφάνεια αφορά την επιλογή των υποθέσεων, τη διενέργεια έρευνας και τον τρόπο με τον οποίο η όλη διαδικασία οργανώνεται στα πλαίσια του Όλαφ. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις ε, διαδικαστικές εγγύησεις, δηλαδή τα δικαιώματα των ερευνόμενων και τη δυνατότητα να έχουμε μία σωστή διαδικασία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα προς τις ε, υποθέσεις που αφορούν εθνικά δικαστήρια έχουμε αποτέλεσμα κατά 30%, δηλαδή έχουμε χαμηλή απόδοση. Θα πρέπει να αυξηθεί λοιπόν η αποδοτικότητά μας, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, δίκες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο και να ευθυγραμμίσουμε τα ε, εθνικά, διοικητικά και δικαιοδοτικά συστήματα έτσι ώστε να στυλιτεύεται η απάτη και να εντοπίζεται σωστά. Αλλά φυσικά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνδράμει ενεργά. Ευχαριστώ και σας καλωσορίσω και εγώ. Πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια του ρόλου σας στο δημοσιονομικό τομέα θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η απάτη μέσα στα πλαίσια των δημοσίων οικονομικών και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θεωρείτε επίσης ότι ο ρόλος του ΟΛΑΦ θα πρέπει να ενισχυθεί. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι η καλύτερη συνεργασία Όλαφ και Επιτροπής Εποπτείας. Πώς βλέπετε το ρόλο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κυρία Λαπάροβα. Ο ενισχυμένος ρόλος του ΟΛΑΦ ε, μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης της απάτης θα ε, σχετίζεται άμεσα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δυστυχώς ε, δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό ο Όλαφ θα πρέπει να συνδράμει όλα τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως προς τα δημόσια οικονομικά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι ο, ο διασυνοριακός ΦΠΑ είναι της τάξης των 150 δις. Το, τα 50 δις αφορούν το εμπόριο τύπου καρουζέλ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταπολεμήσουμε την απάτη που αφορά 10 δις περίπου. Υπάρχουν και οι δημόσιοι διαγωνισμοί καθώς και οι, τα χρηματοοικονομικά μέσα και μηχανισμοί. Υπάρχει ένα σχέδιο που εντάσσεται στη διαδικασία καταπολέμησης της απάτης του Όλαφ. Μπορεί να ενισχυθεί και αν έχω χρόνο θα σας μιλήσω πιο διεξοδικά. Ως προς την Εποπτική Επιτροπή έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τους ελέγχους εξάντε έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικά ε, ανεξαρτησία του Όλαφ και να μπορεί να συνδράμει πραγματικά στην καταπολέμηση. Της απάτης ο συναδελφός Στάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθες, ε, πρώην συνάδελφε. Ποια θα ήταν η στάση σας αν ως μελλοντικός γενικός διευθυντής του Όλαφ ερχόσταν ενώπιον της εξής ε, κατάστασης. Έχετε μια σειρά υποθέσεις που αφορούν τη δική σας χώρα. Γιατί εκεί έχετε και πολιτικό παρελθόν, με πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο, αλλά σε ποιο βαθμό θα μπορούσατε να διατηρήσετε αποστάσεις από πιθανέ υποθέσεις διαφθο... διαφθοράς ή παρατυπιών. Θα τηρούσατε συγκεκριμένη στάση για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από αυτά τα φαινόμενα. Δεύτερον, για την Εποπτική Επιτροπή, συνεχίζω το ερώτημα τη Μαρτίνα. Μεταξύ του πρώην Γενικού Διευθυντή του Όλαφ και τη Επιτροπή αυτή υπήρχε ουσιαστικά ε, έλλειψη ε, συνεργασίας. Δεν υπήρχε βούληση του Γενικού Διευθυντή να ανοιχτεί, στην Επιτροπή αυτή και να δουλέψει και να συνεργαστεί μαζί της με διαφάνεια. Ε, εσείς ε, τι στάση θα τηρήσετε. Ευχαριστώ. Εάν υπάρξουν υποθέσεις που να αφορούν τη χώρα μου, φυσικά και δεν θα εμπλακώ στη λήψη αποφάσεων. Επιτρέψτε όμως γενικά να πω ότι ο Γενικός Διευθυντής της Όλα θα οφείλει να λαμβάνει αποστάσεις από επιμέρους υποθέσεις για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Πρέπει να είναι αμερόληπτος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόθεση που ε, συνδέεται με τη χώρα μου ή με προηγούμενε προηγούμενες θέσεις που κατήχα, ή εγώ ή οποιοδήποτε γενικό διευθυντή, δεν θα πρέπει να εμπλέκεται. Αυτό είναι ασαφέ. Γνωρίζω ε, τις δυσκολίες που υπήρχαν στο παρελθόν ε, στις σχέσεις μεταξύ Γενικού Διευθυντή και Επιτροπής και Εποπτικής Επιτροπής. Συμμετείχα και εγώ σε μια σειρά μακροσπηλών συζητήσεων Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα κανονιστικών, ε, κανονιστικής φύσης. Ε, υπάρχουν ζητήματα που πλέον δεν υφίστανται πλέον πια. Ε, είναι μια νέα εποπτική αρχή, είναι ο κύριος Μούλτα που τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Νομίζω ότι η εποπτική αρχή διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Όλαφ, που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. και βέβαια θα πρέπει ε, να υπάρχει πλήρης ενημέρωση προς την Επιτροπή. Δεν θα εμπλέκεται στην ε, διαδικασία, στην έρευνα, αλλά θα ενημερώνεται. Ο κύριος Δεγιόγκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συνεχίσω στην ίδια άγουσα, γιατί σε ό,τι φορά την πρόσβαση στις πληροφορίες, το θέμα είναι που, τα, που πώς οριοθετούμε αυτή την πρόσβαση το βασικό ζήτημα που υπήρχε στο παρελθόν είναι ε, η πρόσβαση σε πληροφορίες για υποθέσεις που είχαν κλείσει. Και το δεύτερο ερώτημα. Πολλά κράτη-μέλη αναφέρουν σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ο τρόπος ε, που διασφαλίζει τα αποδεκτικά στοιχεία όλα δεν συνάδει με την διαδικασία ε, που υπάρχει αντιστοίχω ε, στα κράτη-μέλη. Τι είδου διαδικαστικά λοιπόν θα ε, μας προσφέρετε για να μην υπάρξουν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Λεγιόν. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι οι διαδικαστικές εγγύησει και το ex monitoring. Αν αποδεχθούμε ότι το δικαστήριο ε, ελέγχει εκ των υστέρων τα όσα κάνει όλα. Οι διαδικασίες που άπτονται των δικαιωμάτων ε, του ερευνόμενου, της πρόσβασης ε, στους φακέλους, σε ένα σωστό χρονοδιάγραμμα, εύλογο χρονοδιάγραμμα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στα άγρια μεσάνυχτα σε ένα γραφείο για να παίρνει αποδεικτικά στοιχεία όλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ε, πρέπει όλα αυτά να τηρούνται ε, παρεγκλήτως για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και υποψίες για τον Όλαφ. Ε, το ένα παράδειγμα είναι ο Όλαφ ε, να ε, εμπλέκεται σε αυτό το, τον εξάντε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνονται εντός, εποπτικής, ε, του Εποπτικού Συμβουλίου, όμως θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες ε, διαδικαστικές εγγυήσεις ε, που θα πλαισιώνουν τις ενέργειες του Όλαφ. Καλησπέρα κύριε Κάλφιν. Θα ήθελα να επιμείνω πιο συγκεκριμένα στο δικαίωμα της υπεράσπασης στα ζητήματα που σας θέσαμε προηγουμένως εξέτασα μία έκθεση ε, του Γαλλικού Κοινοβουλίου πριν από μερικά χρόνια που αφορούσε ακριβώς τον Όλαφ και για τη μεθοδολογία που ακολουθεί. Στη σελίδα 22, για παράδειγμα, μιλούμε ε, για ε, συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρά τις διατάξεις υπάρχουν παραβιάσεις συγκεκριμένων δικαιωμάτων, ε, για το σεβασμό της προσωπικής ζωής και το καθεξής. Αυτό ήταν κάτι το οποίο καταγράφει πολλές φορές ε, και παραβιάζει τα άρθρα ε, της Συνθήκης Διεθνών Δικαιώματα Όλαφ. Οφείλει να διεξάγει δίκαιες έρευνες. Υπάρχουν ζητήματα αδιαφάνειας των ερευνών του Όλαφ εσείς μπορείτε να μας ε, διαβεβαιώσετε ότι αν εκλεγείτε ε, Γενικός Διευθυντής δεν θα υπάρχουν ε, τέτοια φαινόμενα παράνομων διώξεων ή και παράνομων παρεμβάσεων σε εθνικές εισαγγελίες και γιατί, ας πούμε, για τη Γαλλία πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ποινικό αδίκημα, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν θέμα αρχής, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέλω μία συγκεκριμένη δέσμευση. Ah, ah, Ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώ ότι μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι σίγουρα η διατύπωση αυτών ε, των διαδικασιών και η σαφή οριοθέτησή τους. Ε, δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, υπάρχει μία σειρά υποθέσεων ε, στο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δείχνει ότι η έλλειψη εγγυήσεων και εγγύων για τους ερευνόμενους είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα έχει πολλές δυνατότητες που κάποιες φορές ξεπερνούν ε, ε, τα όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για μένα σίγουρα αυτό είναι πραγματική προτεραιότητα και δεσμεύομαι με αυτό. Ο κύριος Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάλφιν, θυμάμαι το καλοκαίρι του 2015 ε, όπου, οπότε και διοργανώσαμε μια ακρόαση που αφορούσε διάφορα ζητήματα που, στα οποία είχε εμπλακεί όλα. Ήταν δύσκολο το θέμα αυτό. Και Μία από τις υποθέσεις που συζητήσαμε ήταν ότι πάνω από το 70% των συστάσεων της, ε, του Εποπτικού Συμβουλίου δεν είχαν εφαρμοστεί από, την, από το Διευθυντικό Συμβούλιο, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μάλιστα ε, ε κάποια στιγμή το Φεβρουάριο του 2012 είχαν ξεκινήσει μέσα σε μία μέρα δεκάδες ε, υποθέσεις. Η διερεύνησή τους δηλαδή. Πώς μπορούμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποφύγουμε στο μέλλον κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόβακοφ. Αυτό σχετίζεται πάλι με το, με το ζήτημα των σχέσεων της ε, Εποπτικής Επιτροπής και του Όλαφ. Μπορώ να επαναλάβω λοιπόν ότι οι, θέσεις αυτές, οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι σχέσεις συνεργασίας. Η Επιτροπική, Εποπτική Επιτροπή ε, είναι το όργανο εκείνο που αποδεικνύει την ανεξαρτησία ε, του Όλαφ. Δεν χωρεί δεν, δεν μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις ε, ε, διαμάχης. Βεβαίως υπήρχαν κάποιες ε, προσωπικές ε, αντιπαραθέσεις, είναι γνωστά αυτά, αλλά τα έχουμε αφήσει πίσω μας πια. Αυτά ε, η Επιπτική Επιτροπή είναι σημαντικό όργανο συλλογής δεδομένων, ανάλυσης επεξεργασίας δεδομένων και όχι απλά μια γραμματεία. Και μάλιστα μπορεί και να ε, ενισχύσει και το έργο της, όπως για παράδειγμα με την εξάντε παρακολούθηση και τις εν γέννη δραστηριότητες του, Αλφα, του Όλαφ. Αυτό λοιπόν πρέπει να εξασφαλιστεί και βάσει και του νέου κανονισμού που έχει τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα. Ακυρώθηκε η πτήση μου από το ε, από το Κάρντιφ. Πολλοί ε, συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην Εποπτική Επιτροπή. Ελπίζουμε όλοι να βελτιωθούν οι σχέσεις. Το ερώτημα μου αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ε, θέσπιση της. Νομίζω ότι θέλουμε όλοι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επικάλυψη του έργου του μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Όλαφ. Αλλά μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποιος ήταν ο ρόλος του Όλαφ στη διερεύνηση και τη δίωξη οικονομικών παρατυπιών ε, όσον αφορά τον ενωσιακό προϋπολογισμό και την ανάκτηση ε, ποσών. Όσον αφορά τις σχέσεις της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Όλαφ, ε, πρόκειται για νομοθετικό έργο που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ελπίζω και νομίζω ότι ο Όλαφ πρέπει να έχει ε, δραστήριο ρόλο στην ε, οριστικοποίηση αυτού του αυτής της σχέσης. Νομίζω ότι μπορούμε να παραδειγματιστούμε από τις εθνικές νομοθεσίες όπου υπάρχουν ε, αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ ε, οικονομικής αστυνομίας ε, και αρχών καταπολέμησης διαφορές, διαφοράς. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το, το πρότυπο πάνω στο οποίο θα βασανούμε. Βεβαίω, δεδομένων των ελλείψεων που ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπάρξουν ζητήματα που θα τα ρυθμίσει ο κανονισμό, Αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το γενικό πλαίσιο δραστηριότητα ε, των δύο φορέων. Βεβαίω και δεν πρέπει να επιτρέπονται επικαλύψει, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να επιτρέπονται και παραθυράκια ε, ή κενά. Ε, ζητήματα στα οποία κανένας από τους δύο οργανισμούς δεν θα έχει την ε, ευθύνη. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει συνεχής ανταλλαγή ροή πληροφοριών και ο Όλαφ πρέπει να επιδιώξει την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ακριβώς διότι οι στόχοι είναι κοινοί και οι λύσεις κοινέ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκρέσλε. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Ποια είναι η εμπειρία σας όσον αφορά την ε, αστυνομική διερεύνηση ε, υποθέσεων. Θέλω να ε, προειδοποιήσω και να πω ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Πρέπει κανείς να έχει και τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη, για να μπορεί κανείς να κατανοήσει και τους καταναγκασμούς υπό τους οποίους βρίσκονται οι φορείς ε, διερεύνησης υποθέσεων. Ε, τι πιστεύετε ότι, ε, ποιος, ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το μέλλον των γραφείων συμψηφισμού και πώς θα εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντή του Όλαφ. Ευχαριστώ. Μιλώ για τις διαδικασίες των γραφείων συμψηφισμού όπου η Κομισιόν Ε, συναντάται με ε, γενικούς διευθυντές προκειμένου να ε, διερευνώνται συγκεκριμένες αποφθέσεις που αφορούν υπαλλήλους της Κομισιόν. Αυτό, αυτό εννοώ. Σε αυτό απαντήστε μου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, πραγματικά δεν έχω ε, ε, εμπειρία σε αστυνομικά ζητήματα, και, αλλά ε, έχω τεθεί και έχω θητεύσει ως επικεφαλής μεγάλων οργανισμών στη χώρα μου και γνωρίζω τα ζητήματα που άπτονται του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εν γέννη ευρωπαϊκών δημοσιονομικών θεμάτων. Ε, και η ακαιρεότητα νομίζω ότι είναι κάτι που, είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Ε, και νομίζω ότι ο Όλαφ έχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη, έχει ε, πολύ έμπειρους υπαλλήλους. Η πρόκληση για μένα δεν είναι να ενισχυθούν οι έρευνες ως αυταξία, αλλά πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία του Όλαφ ε, με όλους τους εμπλεκόμενου φορεί προκειμένου να συλλέγονται πληροφορίε και να αναλύονται. Όσον αφορά την ανεξαρτησία του Όλαφ όταν ε, γίνονται συζητήσει με την Κομισιόν αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο καθήκον τη εποπτική επιτροπή. Ο Όλαφ δεν μπορεί να το κάνει μόνο, μόνος του αυτό. Γι' αυτό έχουμε την, την Εποπτική Επιτροπή πρέπει ο Όλαφ και η, Ευρωπα... και η Εποπτική Επιτροπή να έχουν πλήρη ελευθερία διερεύνησης υποθέσεων όταν απαιτείται. Και όταν γίνονται έρευνες για υπαλλήλους της Κομισιόν πρέπει και πάλι να τηρούνται όλα τα διαδικαστικά εχέγγυα που τηρούνται και στις υπόλοιπες ε, υποθέσεις. Ο κύριος Μπάτσιτς. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Κάλφιν, τον υποψήφιο ενώπιόν μας, που είναι υποψήφιος για μια πολύ σημαντική θέση. Είσαστε ο δεύτερος υποψήφιος και υπάρχει ένα θέμα, ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο μάλλον λύθηκε. Ja, jetzt ist gut. <laughs> Ε, ξέχασα την ερώτησή μου με αυτή τη διακοπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ε, ήθελα να πω είναι ότι είμαι ευγνώμων γιατί φαίνεται ότι ξέρετε πολλά για τον οργανισμό. Έχουν υποβληθεί πολλές ερωτήσεις ήδη. Μία άλλη σημαντική ερώτηση είναι η εξής. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα τρία βασικά καθήκοντα όπου θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές ως προς τις αρμοδιότητες του Όλαφ και πώς μπορεί να αλλάξει η σχέση του Όλαφ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη γιατί πολλά εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι υπεύθυνη νομικά για την δραστηριότητά σας. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτσίτης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι δυνατότητες του εντοπισμού των απατών γιατί υπάρχουν διαφορετικά νομικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε λοιπόν να θέσει υπόψη ένα γενικό ε, μηχανισμό ελέγχου του προϋπολογισμού και επειδή εντασσόμαστε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκείνη θα πρέπει να μας ε, δώσει τα κατάλληλα εχέγγυα για τον εντοπισμό των απατών. Εντασσόμαστε άμεσα στην Επιτροπή και η ερώτησή σας είναι εξίσου σημαντική με την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε. Μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας λοιπόν, ο Όλαφ μαζί με την Εποπτική Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμουν και στους εξάντε ελέγχους. Ο συνάδελφος Πυρίνσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε Κάλφιν η ερώτησή μου έχει ως εξής. Μιλήσατε για τη σημασία επιλογής υποθέσεων και μιλήσατε επίσης για μεγάλες απάτες που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Ξέρετε ότι Υπάρχει μεγάλη ανησυχία φοροαποφυγής, νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία σε αυτό το τομέα. Πιστεύετε ότι ο Όλαφ θα πρέπει να επικαιροποιήσει την επιλογή υποθέσεων έτσι ώστε να μπορεί ο Όλαφ σε επικαιροποιημένε υποθέσεις που δεν απασχολούσαν μέχρι τούδε τον Όλαφ. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που θεωρούνται πιο διεφθαρμένες από άλλες, για να σου το πω έτσι ομά. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Φυσικά ο Όλαφ σας ε, αναφέρεται σε υποθέσεις που αποτελούν μεγάλη επιτυχία σωστές συστάσεις και ούτω καθεξής. Όμως η διαδικασία δημιουργεί ανασφάλεια στο κοινό. Δηλαδή ποιος είναι ο μηχανισμός επιλογής υποθέσεων. Γιατί επιλέγονται ορισμένες υποθέσεις και άλλες όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά μια άλλη πτυχή της προσπάθειας περί διαφάνειας, θα πρέπει να υπάρχουν πιο σαφείς κανόνες. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα νέο κανονισμό για τους εξάντε ελέγχους μέσα στα πλαίσια και του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή η επιλογή των υποθέσεων θα γίνεται από μια νέα μονάδα υπηρεσία μάλλον που θα επιλέγει τις ε, υποθέσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και δεν ε, υποτιμώ τις προσπάθειες εκείνων που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πιο διαφανή κριτήρια για την επιλογή υποθέσεων προς διερεύνηση. Όσο αφορά τις απάτες στο ΦΠΑ και ούτω καθεξής, θα πρέπει να αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Μοσχοβιτσί τώρα ε, ασχολείται με αυτή την πτυχή του ζητήματος που αφορά τις απάτες στο δημόσιο τομέα. Ο κύριος Σαλαφράνκα είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Όπως και στην, ε, στον προηγούμενο υποψήφιο, θα ήθελα και πάλι να χαιρετήσω ένα ενεργό πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει ως εξής. Λάβουμε υπόψη τους πόρους για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρείτε ότι αυτοί οι πόροι επαρκούν γιατί μιλήσατε για τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων και προτεραιότητες δράσεων. Μπορείτε να εμβαθύνετε κάπως τη δράση του Όλαφ. Ε, Επίσης ε, μίλησα και προγενέστερα με τον προηγούμενο υποψήφιο τη σχέση του Όλαφ με τη δική μας Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητά σας έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ μας σε περίπτωση επιλογής σας. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα σας, κύριε Σαλαφράγκα. Αν επαρκούν οι πόροι. Όποιον και να ρωτήσετε από τη διοίκηση θα σας πω όχι. Θα σας πει όχι, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Για τους οικονομικούς πόρους είναι κάτι λιγότερο από 60%, ε, 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο και υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής για άλλα 20 εκατομμύρια που αφορά διάφορες διοικήσεις και εμπλεκόμενους φορείς. Ε, δεν νομίζω ότι οι τρέχουσες συζητήσεις επί του μας επιτρέπουν να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Οι ανακτήσεις ποσών βεβαίων υπερβαίνουν κατά πολύ ε, τον προπολογισμό της Όλαφ. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Όλαφ ε, θα συνεχίσει να εργάζεται με βάση τους οικονομικούς πόρους που δέχεται. Ελπίζουμε και με την ε, σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να παραμείνει το προσωπικό του όλα έχει. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Τα κριτήρια τώρα. Βεβαίως, η εμπειρία μου ε, επί πέντε έτη σε αυτή την Επιτροπή μου δείχνει ότι υπάρχει εξαιρετικά σημαντικό διασύνδεση μεταξύ της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Όλαφ. Γιατί ο Όλαφ έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να ε, διασκεδάζει τις ανησυχίες των πολιτών. Ευθυγραμμίζεται λοιπόν πλήρω ε, και με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ανοιχτοί λοιπόν και εδώ εννοώ διαφάνεια, κανόνε και ούτω καθεξής ίσως χωρίς να μπαίνουμε σε επιμέρους έρευνες για την ερευνητικό μηχανισμό, αλλά οτιδήποτε άλλο, κριτήρια επιλογής ε, υποθέσεων, κριτήρια συστάσεων, σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα και με την Ευρωπαϊκή Συγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να ε, συμφωνηθούν κατόπιν συνένεσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδάλλως πιστεύω ότι ο Όλαφ δεν θα εκπληρώνει ε, το ρόλο του. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πρέπει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε εδώ μαζί μας. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε τον κύριο Κρούβερ να ανέβει στο βήμα. Ε, Καλώ ήρθατε. Αν είστε έτοιμο, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για το γεγονό ότι μου δίνετε το λόγο να σας παρουσιάσω το όραμά μου για τον μελλοντικό ρόλο του Όλαφ και να σας μιλήσω για τα κίνητρά μου και τις εμπειρίες μου, εν συντομία. Θα ξεκινήσω με αυτά τα δεύτερα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το να ηγείται κανείς ενός σύνθετου αξιόπιστου αποτελεσματικού οργανισμού όπως ο Όλαφ χρειάζεται, απαιτεί ε, διευθυντικές και ανθρώπινες δεξιότητες. Δεν μπορεί κανείς να αυτοσχεδιάζει. Πρέπει κανείς να μπορεί να κοιτάζει τα ζητήματα από πολλές ε, ε, οπτικές. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία ε, ξεκίνησε από θέματα ε, διαχείρισης κονδυλίων συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων. Ως πρόεδρος του ομίλου της Αφρικανικής Τράπεζας σχεδίασα και υλοποίησα πολιτικές και στρατηγικές βάση κινδύνου σε διεθνές περιβάλλον και ως εισαγγελέας του ελεγκτικού συνεδρίου ε, υπάρχει κίνδυνος για την ε, κατάχρηση ε, κονδυλίων. Σε μια εβδομάδα θα υποβάλω σχετική έκθεση. Μαζί με την εμπειρία μου έχω και ένα πραγματικό πάθος για την Ευρώπη πραγματικά μου είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, συμμετείχα και στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Γαλλίας ε, και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η ε, Προεδρία του Συμβουλίου να είναι μια συλλογική επιτυχία προς όφελος ε, του κοινού συμφέροντος. Με βάση και τις ιδιότητες και τις θέσεις που κατήχα στο παρελθόν, ε, στην Ινδία και αλλού, ακριβώς αυτούς τους σκοπούς προσπάθησα να πετύχω δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το, με το βιογραφικό μου. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει σύγκληση συμφερόντων γιατί πρέπει κανείς να έχει ε, σημαντική εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό ε, δεν σημαίνει βέβαια ότι ε, μεροληπτώ υπέρ αυτών των σφαιρόντων. ούτε από την άλλη βρίσκομαι ε, τελείως αποκομμένος από όλα αυτά τα πράγματα. Για το μέλλον του όλα αυτά θα ήθελα να σταθώ ε, στις τρεις βασικές προτεραιότητες με βάση την εντολή που θα λάβω. Πρώτον, λογοδοσία, τόλμη και αυτοπεποίθηση. Λογοδοσία λοιπόν, γιατί η ανεξαρτησία και η λογοδοσία είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος. Θα εργαστώ με διαφάνεια, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή μου και από την ε, Εποπτική Επιτροπή του Όλαφ, με τα κράτη-μέλη, τις Εθνικές Αρχές και εσάς και την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και τεράστια ευκαιρία, αν τη διαχειριστούμε σωστά. Δυνατότητα να αυξήσουμε τον αντίκτυπο του Όλαφ, αλλά και να διασφαλίσουμε και την ε, ανάκτηση ποσών, αλλά και την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τόλμη, λοιπόν, να δείξουμε θάρρος ε, και όριμη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να επιλέγουμε υποθέσεις όπου ε, έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή προσταθεμένη αξία, να είμαστε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μας και να διασφαλίζουμε την συνέχεια ε, και να σταθούμε και στην πρόληψη. Κλείνω με την αυτοπεποίθηση. Θέλω να δώσω ε, και να επαναφέρω την αυτοπεποίθηση και την αριστεία, να προσελκύσω ταλέντα, να ε, δημιουργήσω γέφυρες, να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής ε, επανάστασης, αξιοποιώντας το data mining και την ε, τεχνητή νοημοσύνη για να καταπολεμήσω την απάτη και να πείσω τους Ευρωπαίους πολίτες ότι η διαφθορά και η απάτη έχουν περιοριστεί ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και ότι μπορούν να εμπιστεύονται ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κυρίες και κύριοι, για να πετύχουμε σε μία περίοδο προκλήσεων χρειάζομαι τη στήριξη και εμπλοκή σας και μπορείτε πραγματικά να βασίζεστε και στη δική μου βεβαίως στήριξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε πάλι με τον συνάδελφο Ζάβαμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρούγκερ για την ε, εισαγωγή. Οι ερωτήσεις μου θα είναι στα αγγλικά. Πρώτον, Θεωρείτε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου στις έρευνες του Όλαφ. Πιστεύετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει να διαδραματίσει ρόλο και τι σκοπεύετε να κάνετε. Η ΕΚΤ ε, διατηρεί πολλές ε, δυνητικές πληροφορίες για κάποιες υποθέσεις. Δεύτερο θέμα, διαφάνεια. Πώς θα χειριστείτε το θέμα της διαφάνειας ως Γενικός Διευθυντής του Όλεφ. και πώς πιστεύετε ότι εξυπηρετούνται τα δικαιώματα των ερευνομένων ε, όπου ε, η διαφάνεια δυστυχώς ε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πληγεί. Ευχαριστώ. Ξεκινώ με το δεύτερο ερώτημά σας. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να ισορροπήσει κανείς ανάμεσα στη μυστικότητα των ερευνών, την προστασία των πληροφοριοδιωτών, των μαρτύρων κτλ. και την διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα όμω, πρέπει να εξυπηρετούνται και οι δύο στόχοι. Δεν μπορεί να προκρίνει κανείς τον ένα στόχο και να υποβαθμίζει τον άλλον. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση καταλήγουμε ε, σε κακή έρευνα την οποία δεν μπορεί και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω. Όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του Όλαφ, έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας σχετικά με τους συνεργάτες μας, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ ευρύτερη και ε, κοινή χρήση των προφοριών γιατί οι πληροφορίε δεν ανήκουν ούτε στον Όλαφ, ούτε στη Eurojust, ούτε στην Europol, ούτε σε κανέναν άλλον. Αν λοιπόν δεν γίνεται ανταλλαγή των γνώσεων θα χάσουμε ε, αυτόν τον ε, αγώνα εναντίον όσων διαπράττουν απάτες. Ευχαριστώ η κυρία Αγιάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσατε κύριε Κρούγκερ γιατί ε, βρίσκες, ε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της ε, Γαλλικής Γενικής Εισαγγελίας. Ποια είναι η πείρα σας, ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να ε, γίνεται μία έρευνα πιο ενδελεχής. Για παράδειγμα, αν σας καλέσει ε, ένας επίτροπος και σας πει ότι γίνεται απάτη στον τομέα των καπνών, τι θα κάνετε ή τι γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης ε, των δικαιωμάτων των ερευνομένων. Χρειάζεται ένας ε, κώδικας δεοντολογίας. Επίσης υπηρετήσατε στην Τίνιδα κατά την ε, επανάσταση, κατά τη μεγάλη επανάσταση της ε, την Ισίας. Είχατε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που ζήτησαν να γίνει καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Πώς αντιμετωπίσατε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα πλαίσια τη, της θέσης σας στην Αφρικανική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην καριέρα μου είχα πολλές επαφές με τον Όλαφ. Πριν από μία ώρα μάλιστα απάντησα σε αίτημα του Όλαφ που αφορούσε την Κορσική. Βεβαίως για ζητήματα τα οποία, ε, στα οποία δεν μπορώ να επεκταθώ σήμερα, αλλά είναι πολύ ε, ε, ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ότι λίγο πριν πω στην αίθουσα η δουλειά μου είχε να κάνει και πάλι με τον Όλαφ. Εγώ λοιπόν ε, έχω εργαστεί στον εμπορικό ε, κλάδο, όχι στην καταπολέμηση της απάτης, αν και πάντοτε υποστήριζα οι εμπορικές μας συμφωνίες να περιλαμβάνουν ρήτρε καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την υπόθεση Νταλή, αυτό που ήταν πολύ δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι ότι αν ρωτήσετε κάποιον που γνωρίζει την υπόθεση ε, έτσι στο δρόμο που έχει ακούσει για αυτή την υπόθεση δεν, δεν, δεν μπορεί να σας πει ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος ποιος ήταν ο ένοχος γιατί ακριβώς ε, θόλωσαν οι γραμμές κάποια στιγμή και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ε, κανονικά δεν θα έπρεπε ποτέ κανείς να ξεχνά τι καλείται να κάνει, ποιο είναι το καθήκον του. Αν κάποια στιγμή βρεις ενδείξεις ή αποδακτικά στοιχεία τα οποία δεν έπρεπε να είχες βρει, τότε χάνεις την ε, αξιοπιστία σου εσύ ως πρόσωπο αλλά και ως θεσμικό όργανο. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται πάντοτε. Είσαι ε, διοικητικό όργανο, έχεις κάποιους περιορισμούς και κάποια στιγμή πρέπει τις ε, ε, τις πληροφορίες που έχεις συλλέξει να τις παραδώσεις στη δικαιοσύνη. Γιατί οι αρμοδιότητες σου είναι περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει ποτέ να ε, προσπαθείς να ε, συγκεντρώσεις ε, πληροφορίες τις οποίες δεν πρέπει. Για τον Μπέναλή ε, ε, το θέμα είναι περίπλοκο. Η Ισία πριν από 30 χρόνια ήταν μια ευμερούσα χώρα ε, όπου μαζί με την οικονομική ανάπτυξη βεβαίως υπήρχε και σε ένα βαθμό διαφορά. Ε, και όταν δεν αξιοποιούνται βεβαίως σωστά τα δημόσια ε, οικονομικά, τότε καταλήγεις σε τέτοια κατάσταση. Η κυρία Τουμπάζοβα, ευχαριστώ. Ε, η Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντικός εταίρος του Όλαφ. Πώς θα εξασφαλίσετε την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής μας όσον αφορά τις έρευνες του Όλαφ. Και πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά τη ροή προφοριών προς την Επιτροπή μας. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σχετικά με τις ηγετικές σας εικονότητες και την ηγετική σας θέση. Γιατί ο ηγέτης, ο διευθυντή του του Όλαφ θα πρέπει να είναι πραγματικός ηγέτης. Πώς λοιπόν θα δώσετε κίνητρα στους εργαζόμενους ε, του Όλαφ προκειμένου να ε, διεξάγουν τις έρευνες που κάνει ο Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά δεν τίνω να ασκώ κριτική, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά καλύτερα όσον αφορά τη συνεργασία Όλαφ και Επιτροπής Κόντ, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των ερευνών. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια, ή την ποσότητα των πληροφοριών, αλλά και την ποιότητα των πληροφοριών. Και παρακολουθώ πολύ στενά τις εκθέσεις σας και τις συζητήσεις σας για ε, το ΠΙΦ. Νομίζω ότι εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά περιθώρια βελτιώσεων. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά αν θέλει κανείς να χαράσει πολιτική, να προσαρμόζει την πολιτική του, να μετριάζει τον κίνδυνο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν και χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να σκεί πιέσει για να εξασφαλίζεται ότι θα επιτυχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σχετικά με την, ε, τις ηγετικές ικανότητες. Εγώ Είμαι άνθρωπος που δρώ και εργάζομαι συλλογικά. Δίνω κατευθύνσεις, οδηγίες στους υφιστάμενους μας, μου και αυτό θέλω να κάνω και στον Όλαφ. Θέλω να πάω και να πω στους εργαζόμενους του Όλαφ ότι μπορούν να είναι περήφανοι για, τον, για το έργο τους, ότι θα είμαστε μια γροθιά με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και θα εργαστούμε όλοι μαζί. Αλλά χρειάζομαι την συνεργασία σας και την υποστήριξή σας γιατί ζούμε σε εποχή μεγάλων προκλήσεων και αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τον Όλαφ τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε από κοινού την επιτυχία των εργασιών μας. Ο κύριο ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Κρούκερ, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα, Είστε Γάλλος. Φανταστείτε ότι γίνεστε Γενικός Διευθυντής ε, του Όλαφ και στο γραφείο σας κάποια στιγμή καταφθάνουν μια σειρά υποθέσεις ε, που ε, αφορούν Γάλλους υπηκόους, Γάλλους πολίτες. Τι στάση θα τηρήσετε. Θα είστε αμερόληπτος είτε όχι. Δεύτερον, μιλήσατε για το data mining και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσατε ε, να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό το θέμα. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Και τρίτον, για την υπόθεση Ντάλι που μόλις αναφέρθηκε, προκάτοχό σας, επιθανώς ε, προκάτοχό σας, ε, είχα την εντύπωση ότι αυτό ήταν ένα αντικείμενο στο οποίο εξετάζεται έτσι κι ή για, να για την παροχή επαλλαγή. Ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα για τη Γαλλία. Πραγματικά θα είμαι αμερόληπτος. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι και με τη σημερινή ιδιότητά μου δεν έχω πολλούς φίλους ε, στη Γαλλία και είχα δυνατότητα να κάνω αυτή τη δουλειά γιατί είχα περάσει μια δεκαετία στο εξωτερικό. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει ανεξαρτησία και αμεροληψία, καθώς και λογοδοσία. Γι' αυτό και επέμεινα τόσο στη λογοδοσία. Δεν θα είμαι βέβαια μοναχικός ε, καβαλάρης, θα είμαι εδώ μαζί σας ενώπιον ε, των ε, εκπροσώπων δηλαδή, δηλαδή των πολιτών θα είμαι εξαιρετικά διαφανής ε, και αμερόληπτος. Και δεν έχω καμία αφιβολία ότι θα συνεχίσω να είμαι το ίδιο αμερόληπτος όσο είμαι σήμερα έναντι των γαλλικών αρχών. Ε, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι κέρια σημασία θέμα. Αν είχα χρόνο να αναφέρω και ένα τέταρτο στοιχείο των τριών που ανέφερε προηγουμένω, θα ήταν τα δεδομένα. Έχω ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα στο Ελληνικό Συνέδριο στη Γαλλία. Είναι ένα πραγματικό αγώνα. Μέσα σε μερικά. αγώνα ταχύτητα εννοώ. Μέσα σε μερικά λεπτά μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με την απάτη καρουζέλ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε τεθειμένοι να κάνουμε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ιδίω ό,τι αφορά του φόρου. Αν δεν έχουμε δυνατότητα λοιπόν να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα με τεχνολογίε εχμή και τα πιο αποτελεσματικά μέσα, είμαστε χαμένοι από χέρι. Εδώ ο υπολογιστής κέρδισε τον Γκασπάροφ στο σκάκι και πλέον έχουμε μια νέα γενιά υπολογιστών που μέσα σε μισή ώρα από εκεί που δεν ήξεραν καθόλου τους κανόνες τώρα κερδίζουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, όλα τα μέσα που μπορούμε να ε, αποκτήσουμε γιατί πρέπει να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες φυσικά στις έρευνές μας αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, υπέρ ή κατά. Ε, αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει κανεί να έχει μια εξορροπημένη ε, προσέγγιση. Δεν γίνεται να πάμε μόνο λοιπόν επιθετικά. Πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη ε, προκειμένου η υπόθεση που θα στείλουμε τελικά στη δικαιοσύνη θα ευσταθεί και δεν θα πρέπει να ξανακάνει η δικαιοσύνη την ίδια δουλειά. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να συνεχίσω σε ό,τι αφορά την πρόληψη ε, των συγκρούσεων συμφερόντων. Φυσικά και όλα θα έχει ε, αρμοδιότητα και ευθύνη έναντι των κρατών μελών και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, υποθέσεις εντός της Κομισιόν. Ποιες είναι οι σχέσεις, θεωρείτε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, πολλά έχουν υποθεί για την ε, ε, συλλογή δεδομένων και τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια για τα κράτη-μέλη και τους ε, εισαγγελείς. Αυτό κάποιες φορές είναι προβληματικό. Θεωρείτε ότι μπορούν να υπάρχουν και εξωτερικοί έλεγχοι ή διαδικαστικές εγγυήσεις ή οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται εσωτερικά. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και τι διαδικαστικέ εγγύησει, ευχαριστώ για τα ερωτήματά σα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι έχει δύο σκέλη η Όλαφ, ε, πολιτική πρόληψη και διερεύνηση. Πρόκειται για ξεχωριστά σκέλη, αλλά υπάρχει άλλη αλληλεπίδραση. Γιατί αν υπάρχει σωστή πρόληψη, τότε αυτό διευκολύνει και το έργο των ερευνητών και το αντίστροφο. Βέβαια, αν κανείς ενεργεί υπό την ιδιότητα του ερευνητή, έχει πλήρη ανεξαρτησία. Αυτό ισχύει από ε, την αρχή της ύπαρξης του Όλαφ, το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να είναι κανείς αρκετά ευφυής για να ακούει να είναι εταίρος ε, της πολιτικής, αλλά παράλληλα και να μην επηρεάζεται εύκολα ε, κατά τη διάρκεια των ερευνών για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Για την συλλογή δεδομένων και η προσθέμενη αξία των εκθέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέλημα για μένα. Ελπίζω όταν αναθεωρήσετε τον κανονισμό του 13 για τον Όλαφ, θα βρείτε έναν τρόπο, ελπίζω, ε, για να ενισχύσετε αυτή την πτυχή. δεν είναι δυνατόν όταν γίνεται σωστά μια ε, τέτοια διαδικασία, ορισμένα κράτη-μέλη ε, να ασκούν η εισαγγελικη εισαγγελική δίωξη, ενώ άλλα κράτη-μέλη να ξαναρχίζουν την έρευνα. Και έτσι χάνεται πολλή χρόνο. Κάποιε φορέ υπάρχει ακόμα και παραγραφή του αδικήματο. Το 1 τέταρτο των ε, συστάσεων του Όλαφ είναι ε, δικαστικής και το 1 τέταρτο αυτών των συστάσεων οδηγεί σε δίωξη. Δεν μιλώ καν για τι κυρώσει, γιατί τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα και δεν υπάρχουν στα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να αλλάξουμε άρδιν αυτή την εικόνα. Ο συνάδελφος Ζάκ. Καλώς σας βράδυ κύριε Κρούγκερ ε, και καλώς ορίσατε. Ως προς την ανεξαρτησία του ΟΛΑΦ, ε, όταν δούμε τη θεωρία, βλέπουμε ότι ο Όλαφ θεωρείται ένα ανεξάρτητο όργανο με βάση τα άρθρα 3, 4, 5 του κανονισμού 99 και 11 και 12 του κανονισμού 1073 και 1074. Τα πράγματα όμως στην πράξη είναι λίγο πιο περίπλοκα. Η Γαλλική Γερουσία εξέδωσε ένα έγγραφο ως προς τους ανεξάρτητους οργανισμούς στη Γαλλία. Έγινε όμως λόγος και για τον Όλαφ και η έκθεση αυτή θεώρησε ότι ο Όλαφ δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός με βάση τα γαλλικά κριτήρια. Άρα θα πρέπει να δούμε καταρχήν ποιες θα είναι οι σχέσεις του, της Εποπτικής Επιτροπής και του Όλαφ, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του οργανισμού. Φαίνεται ότι απέχουμε πόρο από αυτή την κατάσταση αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα της Εποπτικής Επιτροπής. Άρα η οι όροι ήταν αρκετά έντονοι, διότι ο προκάτοχός σας ε, ε, κατηγόρησε την ε, Επιτροπή ότι δηλαδή το, η έκθεσή της ε, μεροληπτούσε. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να απαλύνετε αυτή την κατάσταση και για να μην υπάρχει η υποψία περί μεροληψίας και έλλειψης ανεξαρτησίας του ΟΛΑΦ. Κάτι το οποίο στοιχίζει χρήματα στον ε, Ευρωπαίο φορολογούμενο και από όσο γνωρίζετε υπάρχει και μια οδηγία σε σχέση με τους ελεγκτές που τώρα έχει στην ουσία αφοπλιστεί. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ως προς την Εποπτική Επιτροπή θα ήθελα πράγματι να υπάρχει μια καρποφόρα συνεργασία με τον Όλαφ. Ο πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής παρακολούθησε όλες τις ακροάσεις ε, στις οποίες συμμετείχα και πάντα ήμουνα πολύ ειλικρινής. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι της ε, γάτας και του ποντικού υπεξερώντας πληροφορίες και κάνοντας παράλογες προσφυγές της νομικές υπηρεσίας. Νομίζω ότι πρόκειται για έναν θεματοφύλακα της ανεξαρτησίας, περί ανεξαρτησίας. Αυτό ακριβώς ορίζει ο κανονισμός του 73 και θα ήθελα να ε, υπάρξει μια διαδικασία εργασίας και συνεργασίας με την Εποπτική Επιτροπή. Ως προς την ανεξαρτησία, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο ε, ξεχωριστές αρχές. Η μία είναι ανεξάρτητη, η άλλη όχι. Υπάρχει μία διάδραση μεταξύ του κόσμου της έρευνας και του κόσμου της πρόληψης. Ο κόσμος της έρευνας θα είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Τώρα, ως προς την πρόληψη και την ασφάλεια διαδικασιών για να αποφύγουμε την ε, απάτη θα πρέπει να πρόκειται για, ένα, να πρόκειται για έναν συλλογικό μηχανισμό, Νόβακοφ. Ευχαριστώ. Κύριε Κρουγκέρ, αύριο ο πρόεδρος Μακρόν στην Ολομέλεια θα μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης μίλησε για βαθιές ε, μεταρρυθμίσεις στην ε, απαρχή της θητείας του. Εσείς νομίζετε ότι θα μπορέσετε να ε, επηρεάσετε αυτή την πορεία εάν χρηστείτε γενικός διευθυντής του Όλαφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τον Όλαφ, η ατζέντα είναι πολύ φορτωμένη. Έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε δύο χρόνια, τον, ε, το κανονιστικό πλαίσιο σε δύο μήνες. Ο Ευρωπαίος πολίτης θεωρεί ότι η απάτη είναι υψηλότερη από ότι δέκα χρόνια πριν. Υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία δεν μας φέρνει καλά νέα ως προς τον Όλαφ. Γι' αυτό νομίζω ότι ε, η ατζέντα είναι πολύ φορτωμένη. Ξέρω τι μπορώ να κάνω εάν αναλάβω αυτό το χρήσμα και αυτό αφορά και την πανεκκίνηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος γενικότερα. Σε σχέση με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρόεδρος ε, Μακρόν έχει ασχοληθεί επί του θέματος και νομίζω ότι θα υπάρξει μία καρποφόρα συνεργασία ως προς την ε, δημοσιονομική διαδικασία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ε, τεχνητή νοημοσύνη προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την συνεισφορά σας. Σε σχέση με την ε, Εποπτική Επιτροπή θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η αγαστή συνεργασία, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Ποιο ήταν το πιο ακαθόδες πρόβλημα. Γιατί υπήρξε αυτή η, η, η κακή σχέση με την Εποπτική Επιτροπή σε σχέση με τον ΠΟΕ θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επικάλυψη αυτού του οργανισμού με το έργο ε, του Όλαφ. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει επικάλυψη. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η επικάλυψη βεβαίως απασχολεί τη, τη συζήτηση. Αν και δεν είναι το κύριο θέμα, κατά τη γνώμη μου. Από την εμπειρία μου, στη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων, προτού παραδώσει κανείς την υπόθεση στη δικαιοσύνη, πρέπει να συλλέξει όρημα, επαρκή στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί αν δαπανίσεις υπερβολικά πολύ χρόνο, παραδίδεις την υπόθεση υπερβολικά αργά στη δικαιοσύνη, ε, με πολλές διαδικασίες, ε, ενώ αν από την άλλη μεριά ε, προχωρήσεις πάρα πολύ γρήγορα, θα έχεις μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα απασχολείται με υποθέσεις που δεν είναι όριμες όπως είναι η διασυνοριακή χρηματοδότηση της δημοκρατίας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εμπειρία, πείρα ε, όσον αφορά τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχουν και περιπτώσει όπου και εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό, αυτό θα είναι ε, αρκετά δύσκολο ε, προκειμένου να ε, εξευρεθεί η σωστή ισορροπία. Για το άλλο ζήτημα που θέσατε. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πτυχέ. Πρώτον υπάρχει η έλλειψη πληροφοριών, για τη διαφάνεια δηλαδή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά και κάποια από τα αιτήματα της Εποπτικής Επιτροπής ήταν υπερβολικά ε, στο παρελθόν. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο τρόπος ε, για να πετύχουμε είναι να προστατεύει κανείς και να υπερασπίζεται τα δικά του ε, καθήκοντα. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λειτουργεί πολύ σωστά δεν βρίσκονται ε, προβλήματα από την, Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλήματα που ε, στο τέλος τα εντοπίζει όμως όλα. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό, γι' αυτό το γεγονός ότι πολλά προγράμματα ολοκληρώνονται ε, χωρίς προβλήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν καλείται να διερευνήσει τα προγράμματα αυτά Όλαφ τελικά εντοπίζει παρατυπίες. Πιστεύετε ότι Πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρξουν βελτιώσεις σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών με την Κομισιόν ε, για τα προγράμματα και πώς θα καταστήσετε την όλη αυτή διαδικασία πιο ορατή, πιο διαφανή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ εξεπλάγην στην αρχή της υποψηφιότητάς μου για τον Όλοφ από ε, τον αριθμό των ε, υποθέσεων όπου υπήρχε μεγάλη διαφορά ως προς τις συστάσεις και ως προς την εκπλε... Ε, εκτέλεση, την υλοποίηση των συστάσεων. Και πηγή αυτών των διαφορών είναι οι διαφορές που υπάρχουν στις διαδικασίες. Εγώ δεν πρόκειται να κλείσω ποτέ μια υπόθεση αν δεν βεβαιωθώ ότι έχω καταλάβει τη θέση εκείνων που έχω ερευνήσει και ότι εκείνοι έχουν καταλάβει τη δική μου θέση. Διότι αν καταλήξεις σε έλεγχο, σε έκθεση, σε, σε, σύνταξη έκθεσης που περιλαμβάνουν ε, σφάλματα ε, από την αρχή, ε, τότε βεβαίως θα καταλήξεις και σε λανθασμένα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι πολλά από τα προβλήματα σε μεταγενέστερο στάδιο μπορούν να επιλύονται αν υπάρχει σωστός ε, και ο κατάλληλος διάλογος ε, στις ε, αρχικές φάσεις της διερεύνησης των υποθέσεων. Ο κύριος Μπάτσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι κυριότερος στόχος μας και κυριότερος στόχος δικό σας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι υποθέσεις απάτης θα μειωθούν στο μέλλον. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο απαιτείται στενότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 κράτη-μέλη. Μάλλον σύντομα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 27. Και σε κάθε κράτος μέλος, κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται εκλογές, αλλάζουν πολιτικοί, αλλάζουν κυβερνήσεις και αλλάζουν και οι πολιτικές μαζί με τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε στενότερη συνεργασία του Όλαφ με τις κυβερνήσεις και τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των κρατών μελών, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη σε σχέση με την πρόληψη αλλά και την ε, επίτευξη συμφωνιών που θα επιτρέπουν στον Όλαφ να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Και πιστεύετε ότι είναι δύσκολο το καθήκον αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτό το καθήκον και πολύ δύσκολο και για μένα να το εκπληρώσω. Αυτό είναι βέβαιο. Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη ε, στα έσοδα και τις δαπάνες είναι πραγματικά πολύ σημαντικός και βλέπουμε ότι έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που οι μονάδες ε, συντονισμού για τη διαφθορά στα κράτη-μέλη δεν είναι τόσο δραστήρια. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε. Εγώ θέλω να αλλάξω. Πρέπει ε, να διαμορφώσουμε ένα πραγματικό δίκτυο ε, εντός του οποίου θα ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές για να γνωρίζουμε ότι αν υπάρχει ένα ζήτημα εφαρμογής των διαρευνητικών αρμοδιοτήτων της Όλαφ ή που έχει βρεθεί μία λύση ε, σε μία χώρα, να μπορούμε να βρίσκουμε αυτές τις λύσεις σε οποιαδήποτε χώρα. Κάποια κρατημέλη έχουν ε, χαράξει μια εξαιρετική πορεία για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και εμείς δεν το εξετάζουμε ολοκληρωμένα, εξετάζουμε με μονομένες περιπτώσεις. χάνοντας ε, την ευρύτερη εικόνα και την πορεία που έχει σημειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ εκ μέρους του ΕΛΚ τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η εμπειρία σας όσον αφορά τις αστυνομικές έρευνες. Δεύτερον, τι πιστεύετε τις διαδικασίες γραφείων συμψηφισμού. Δηλαδή, τις μηνιαίες συζητήσεις μεταξύ Κομισιών και Γενικής Γραμματείας σχετικά με τις υποθέσεις όλα που αφορούν υπαλλήλου της Κομισιόν. Γιατί εδώ τίθεται το θέμα της ανεξαρτησίας του οργανισμού. Και τρίτον, ε, υποστηρίζετε η υποψηφιότητά σας από τη γαλλική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. I start with the last question. Ξεκινώ με το τελευταίο ερώτημά σας. Σαφώς και υποστηρίζετε, ελπίζω τουλάχιστον, αλλά ε, η υποψηφιότητά μου δεν είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης της γαλλικής κυβέρνησης. Εγώ έθεσα την υποψηφιότητα. Βρισκόμουν σε μια βαρετή συνάντηση και κοιτούσα το κινητό μου και είδα ότι υπάρχει μια θέση που ανταποκρίνεται ακριβώς ε, ε, στι δεξιότητέ μου και λέω γιατί όχι, να θέσω ψηφιότητα. Αυτό ήταν η αρχή αυτή τη περιπέτειας. Για ε, τα γραφεία συμψηφισμού Clearing House αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Μπορεί κανείς να το εξετάσει ως επιρροή των διερευνητικών αρμοδιοτήτων. Από την άλλη όμως διασφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων το γεγονό ότι βρισκόμαστε στην ίδια αίθουσα δεν σημαίνει ούτε ότι συμφωνούμε, ούτε ότι βγαίνοντα θα ξεχάσουμε τα καθήκοντά μας και την εντολή μας. Έχω μακρά εμπειρία με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και βλέπω ότι είτε οι ερευνητές ξεχνούν τα καθήκοντά τους και δεν διερευνούν ή από την άλλη, αντίθετα, ψάχνουν να βρουν το οτιδήποτε για να φτιάξουν το φάκελο. Πρέπει λοιπόν εμείς να παραμείνουμε ήρεμοι και να συνεχίσουμε την έρευνα όπως κάνουμε με οποιαδήποτε άλλη έρευνα. Και βοηθάει το clearing house αυτή τη διαδικασία. Τώρα, στις αστυνομικές ε, έρευνες έχω μία διτή εμπειρία. Αφενός, ε, συνεργασία με τις δικαστικές ε, αρχές στη Γαλλία, και σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Έτσι είχα έρθει δηλαδή σε επαφή με, τους, ε, με την αστυνομική δίωξη, την αστυνομική έρευνα, μέσω του δικαστικού συστήματος δηλαδή. Αλλά και προέρχομαι, ε, μάλλον στο κατά το παρελθόν ήλεγχα την ε, αστυνομία, έτσι ξεκίνησα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση. Χαιρόμαστε για την παρουσίαση. σας. ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πρέπει να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Wir haben den Herrn Litzke als letzten. Kommt genau, in front of the door. Thank you so much. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν, αν θέλετε, αν είστε έτοιμος. Παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου σε περίπτωση που με επιλέξετε ως μελλοντικό Γενικό Διευθυντή του Όλαφ. Πρώτον, ποιος είναι, ποια, είναι η σχέση του Όλαφ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, καθορίζεται στον ε, σχετικό κανονισμό ε, στους σχετικούς κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τον Όλαφ. Δεν υπάρχουν επικαλύψεις, συμπληρωματικός είναι ο ρόλος τα οικονομικά εγκλήματα θα διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Συγγελία. Θα αλλάξει ο, ο ρόλος του Όλαφ. Θα επικεντρώνεται σε διοικητικές διαδικασίες και έρευνες που θα αφορούν και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κεντρικές δαπάνες καθώς και το ΦΠΑ ε, όπου οι υποθέσεις δεν είναι διασυνοριακές και αφορούν λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο του Όλαφ στο μέλλον, εξ όσων καταλαβαίνω, θα αφορά περισσότερο τη συνοχή πολιτικής, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον έγκαιρο, την έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη και τη συλλογή πληροφοριών. Το άρθρο 1, παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκαθαρίζει ότι ε, πρόκειται για συνεργασία, συντονισμό και υποστήριξη Τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό λοιπόν, μόνο σαφήνεια. Αυτό από την άλλη πλευρά για μένα, σε περίπτωση που εκλεγώ ω Γενικό Διευθυντή του Όλαφ, σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να έχω κατά νου το, τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι αλλαγές στο προσωπικό του Όλαφ. Το προσωπικό, εξ όσων γνωρίζω και έχω συνεργαστεί με πολλούς από το προσωπικό του Όλαφ, είναι εξαιρετικό και είναι πολύ περήφανο για το γεγονό ότι ε, εκτελεί και εισαγγελικές ε, δραστηριότητες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι στο μέλλον ε, ενδέχεται να ε, προκληθεί φόβος από τις εξελίξεις που έχουν. Για να αποφευθεί κάτι τέτοιο, εγώ ως μελλοντικός διευθυντής του οργανισμού, αν με εκλέξετε, θα πρέπει να προσφέρω στο προσωπικό ένα νέο νόημα στη δουλειά τους που θα που μπορεί να σημαίνει μόνο την ε, ανάπτυξη και την προαγωγή ε, στον χώρο εργασίας, για παράδειγμα με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Συγγελία και με περισσότερη υποστήριξη από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι μπορώ να κάνω ακριβώς για να επιτύχω αυτό το στόχο ε, ως άτομο, ως πρόσωπο. Ο ρόλος μου θα είναι να γεφυρώσω την λειτουργία του Όλαφ στη νέα εποχή με ε, μετριοπάθεια και με ηγετικές ικανότητες. Μετριοπάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό που με διακρίνει ε, ε, σε όλες τις θέσεις που κατήχα στην ζωή μου και στον, στην, στον ΠΟΗ και στον, στον ΟΗΕ όπου ακριβώς αυτό κάνουμε ε, γεφυρώνουμε ε, τη μετάβαση ε, από παλιές ηγεσίες σε νεότερες. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που αφορά και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το δικό σας. Καταλαβαίνω ότι η σχέση δεν ήταν πάντοτε η καλύτερη με τον Όλαφ, Αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, όμως σε, στο μέλλον η εταιρική σχέση μεταξύ ε, του Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και με την Εποπτική Επιτροπή ε, και με την δική σας Επιτροπή, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Τι άλλο κομίζω. λένε για μένα ότι είμαι ιδιαίτερα χαρισμητικός, μπορώ να, να ενθαρρύνω και μπορώ να αξιοποιήσω δίκτυα και το, η θέση του Γενικού Διευθυντή του Όλαφ μπορεί να είναι πολύ μοναχική κάποιες φορές και καταλαβαίνω ε, ότι έτσι ήταν στο μέλλον. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να συνεργάζεται και με τους διευθυντές και με το προσωπικό, με το προσωπικό της Κομισιόν, με τη δική σας Επιτροπή, με το Συμβούλιο και εγώ, εμένα η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή όποτε μου ζητείτε η συμβουλή μου και όπου μπορώ να μάθω. Και είμαι πολύ σαφής σε αυτό, ότι θα χρειαστεί και εγώ να μάθω πολλά. Τι άλλο κομίζω. Εγώ ήμουν επικεφαλής ε, ερευνητής σε πολυεθνικούς οργανισμούς με 194 κράτη-μέλη όπου οι διαφορές μεταξύ χωρών, πολιτισμών, ε, πεπιθήσεων, ε, απόψεων είναι τεράστιες και μπορούν να γεφυρώνονται κανείς, να, να γεφυρώνονται μόνο με τέτοιες ήπιες και μετροπι, μετριοπαθείς κινήσεις. Επίσης, ε, πολλές φορές τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν να προστατευτούν τα δικαιώματα των ερευνομένων. Εγώ το έχω κάνει αυτό, γιατί ως δικαστής ε, που έχω υπάρξει κάνει κανείς ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ ε, της αγωγής και των ε, εναγωμένων. Είμαι και πατέρας. Έχω ε, ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή μου ε, εμπειρία. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ε, έχω εργαστεί 15 χρόνια για τον ΟΗΕ και τους εξειδικευμένους οργανισμούς του. Σήμερα οργάζομαι για ζητήματα ηθικής στην Ιεμένη, στη Συρία. Ό,τι και αν σκεφτείτε έχουμε παρουσία. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχω συμπροεδρεύσει ε, πριν από 10 χρόνια περίπου ε, την Task Force έρευνας ε, την κοινή Task Force ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο. Επίσης δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων και είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριο Σάββαμα. ξεκινάει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, για, τις, για τα στοιχεία που μας δώσατε. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο και ποιος θα είναι αυτό όσον αφορά τις έρευνες του Όλαφ. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Τι θα κάνετε στο θέμα αυτό. Και δεύτερο, διαφάνεια πώς θα χειριστείτε το θέμα συνολικά της διαφάνειας ως Γενικός Διευθυντής του Όλαφ και τι πιστεύετε για τα δικαιώματα των ερευνομένων και την προστασία τους. Πώς πιστεύετε και τι πιστεύετε ε, σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των ερευνομένων σε, ένα, σε έναν Όλαφ που μέχρι στιγμής ε, δεν ήταν πάντοτε, δεν χαρακτηριζόταν πάντοτε από απόλυτη διαφάνεια. Το θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου ε, είναι ένα ουσιώδες ε, ζήτημα για τον Όλαφ με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Πιστεύω ότι θα υπάρχει αγαστή συνεργασία και με το ελεγκτικό συνέδριο και στα Ηνωμένα Έθνη και στον ε, ΠΟΕ είδα ότι μόνο με τη συνεργασία επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Όταν μιλάμε για δίκτυα, υποστήριξη και αλληλοσυμπληρούμενες ε, ε αλληλοσυμπληρούμενους οργανισμούς μπορώ να πω ότι πρώτη στο στόχο είναι η συνεργασία με το ελεγκτικό. Τι σημαίνει διαφάνεια. Διαφάνεια σημαίνει ε, λογοδοσία. Θα πρέπει να δούμε πόσο ε, διακατέχεται από διαφάνεια η εργασία του Όλαφ. Υπάρχουν βεβαίως και θέματα απορρίτου. Όμως θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία του Όλαφ έναντι της Εποπτικής Επιτροπής και της δικής σας Επιτροπής. Και ως προς τα ατομικά δικαιώματα κατανοώ το ερώτημά σας σε σχέση με διαδικαστικά εχέγγυα και εγγυήσεις και θα συνεργαστώ μαζί σας και σε αυτό. Η κυρία Γιάλα. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Μίτσκε, τον τελευταίο μας υποψήφιο. Ε, βλέπω ότι δεν κατανοείτε την Ισπανική παρόλο που συμμετείχατε στα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, μάθατε για αυτή τη θέση και γιατί ε, εκφράζεται ενδιαφέρον να επιστρέψετε στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε πραγματικό ενδιαφέρον πέρα από το επαγγελματικό ιδιαίτερα όταν μιλήσατε για σύγκρουση, για βασικές ε, συγκρούσεις, ιδιαίτερα στη Συρία, Πέδιο και είδαμε τι έγινε και με τον οργανισμό ανοικοδόμησης. Ας μην επεκταθώ επί του θέματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια, ποιες ήταν οι επιτυχίες σας στην ε, καταπολέμηση της απάτες, της απάτες και τι κάνατε στα πλαίσια των ε, Ηνωμένων Εθνών για να καταπολεμήσετε την απάτη και ιδιαίτερα στις σχέσεις ε, με εμπλεκόμενους φορείς όπως είμαστε και εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του ε, των Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελα να μας πείτε αν γνωρίζετε προσωπικά την κυρία Γεωργίβα. Ε, θα απαντήσω στα αγγλικά. Καταρχήν πώς έμαθα για αυτή τη θέση. Έχω ένα πολύ ε, καλό δίκτυο και ο, η θέση του Γενικού Διευθυντή στον ΟΛΑΦ είναι η πιο ε, προεξέχουσα, προεξάρχουσα θέση για την καταπολέμηση της απάτης πέρα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή είναι η έκτη συνέντευξη που, στην οποία συμμετέχω και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, μεγάλες επιτυχίες. Ως ερευνητής έμαθα ότι πρέπει κανείς να είναι πολύ υπομονετικός. Δεν θα σας πω ότι κατάφερα, ε, ότι είχαμε τεράστιες επιτυχίες και ούτω καθεξής. Ε, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν στο Κωσυφοπέδιο όταν ε, σε ένα διαγωνισμό, όταν ακυρώθηκε ένας διαγωνισμός για ένα ηλεκτρικό δίκτυο. Ήταν της τάξης των 5 εκατομμυρίων συμμετείχαν και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μάθει να εργάζομαι με περιορισμένους ε, πόρους, δηλαδή να θεωρώ ότι όταν κερδίσουμε 50.000 δολάρια ή 100.000 δολάρια, ενώπιον ενός δικαστηρίου αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Αν μπορεί κανείς να επηρεάσει ένα σύστημα έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα ε, ε, ε, δημοσίων προμηθειών, τότε αυτό αποτελεί επιτυχία. Δεν θέλω να το, να το παίξω σε ρήφης ή τιμωρός. Η αντιμετώπιση της απάτης, η μεγαλύτερη μου επιτυχία, ήταν η ακύρωση ενός διαγωνισμού στο Κωσυφοπέδιο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λαμπάιωβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το βιογραφικό σας είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είπατε κι εσείς ε, από την άλλη ότι δεν έχετε μεγάλη ε, πείρα από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και ε, σχετικούς μεγάλους οργανισμούς. Τι έχετε να μας προσφέρετε ως αντιστάθισμα της έλλειψης εμπειρίας αυτής και πιο τεχνικό σκέλος τώρα υπάρχει ένα benchmark 12 μηνών για τη διάρκεια των ερευνών στον Όλαφ ενώ ο προηγούμενος Γενικός Ευθυντής θέσπισε ένα ε, σημείο αναφοράς 20 μηνών σε ό,τι τις έρευνες. Ποια είναι η δική σας θέση ως προς τη διάρκεια των ερευνών, γιατί μεγάλος αριθμός των ερευνών υπερβαίνουν τους 12 μηνών, ε, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα ε, συρρυκνωθεί το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα είναι κάπως προκλητική απάντησή μου. κανένα μάνατσερ δεν μπορεί να χειριστεί πάνω από 8 με 10 άτομα υφισταμένους. Όταν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την ηγεσία, ε, το θέμα είναι ποιους ε, ακριβώς... Ποιον υγείσαι, ποια είναι αυτά τα 8-10 άτομα που είναι άμεσα εφισταμενοί σου. Ε, μιλήσετε με τους ε, συναδέλφους μου ε, στον ΠΟΗ, που είναι μεγάλος ε, Παγκόσμιο οργανισμός, δεν είναι ο μεγαλύτερος βέβαια, ο ΙΕ είναι μεγαλύτερος, θα δείτε ότι έχω αυτές τις δυνατότητες και πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν μπορεί κανείς να πει κάθε φορά έχω ήδη εμπειρία και θα συνεχίσω στην επεβατημένη. Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά το θέλω. Δεύτερον, για τη διάρκεια. Καμία ερευνητική αρχή από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει που να μην δυσκολεύεται με τα χρονοδιαγράμματα και τα σημεία αναφορά στα benchmarks γιατί υπάρχει και η επιδίωξη της αριστείας ε, και το καθήκον, ότι πρέπει δηλαδή κανείς να κάνει τη δουλειά του σωστά, ακόμα και να του πάρει μια μέρα παραπάνω. Μετά, είμαι πεπισμένος ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η στενή συνεργασία με τον Όλαφ θα συνδράμουν περαιτέρω στην προσπάθειά μας να φτάνουμε μέχρι τέλους ε, στις έρευνές μας. Λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα είπε ο κύριος Σάβαρμα, αν ε, έχουμε πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών ε, με την εισαγγελία, τότε θα διατηρήσουμε, θα σεβαστούμε και το benchmark αυτό και θα πέσει η μέση διάρκεια των ερευνών. Ο κύριος Στάς, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Με ενδιαφέρει αυτό που είπατε για την εμπειρία σας στο κοσμοπαίδιο. πιο συγκεκριμένα για, ε, για το αεροδρόμιο ε, της ε, Πρίστινα ε, και, για την εταιρεία ηλεκτρισμού, την ΚΕΚ. Ήταν μια έρευνα απάτη, απάτης, τι ακριβώς χαρακτήρα είχε και ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος. Πράγματι υπήρχε, υπήρξε έλεγχος που επεσήμανε ορισμένες πιθανές ε, παρατυπίες και ως εκ τούτου ήταν η πρώτη συνεργασία εκείνη τη στιγμή υπό τον Γενικό Γραμματέα Εποπτείας που ε, δημιούργησε την μια ερευνητική task force. Ένα θεσμικό όργανο με επικεφαλής του, στον ΟΗΕ και επικεφαλής της Βρυξέλλες τον κύριο Μπρούνερ και Είχαμε και δύο επιχειρησιακούς επικεφαλείς. Εγώ ήμουν αναπληρωτής επικεφαλής από πλευράς ε, ΟΗΕ. Ξέραμε όμως πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα, γιατί δεν είχαμε τις ίδιες διαδικαστι... τα ίδια διαδικαστικά ειχέγγυα. Οπότε έχω αυτή την εμπειρία ε, επειδή υπήρχε στενή συνεργασία. Ήταν δύσκολο βέβαια αυτό το εγχείρημα, δύσκολη και η συνεργασία μας. Υπήρχαν ορισμένες τριβές. Είχαμε 15 έρευνε, 12 έφτασαν σε δίωξη από διεθνή εισαγγελέα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, γιατί ήταν επικράτεια την οποία διαχειριζόταν ε, ο ΟΗΕ. Εγώ λοιπόν, ως επικεφαλής για τη στιγμή, άσκησα ε, διοικητικές ε, αρμοδιότητες σε αυτή την επικράτεια. Και αυτό φυσικά είχε τεράστιες, ε, τεράστια ευθύνη. Δεν τα έκανα όλα σωστά, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία μας ήταν ότι βρήκαμε τους συνδέσμους μεταξύ της διαφθοράς και άλλων αντικειμάτων που διερευνώνταν εκείνη την περίοδο στο Κωσοφοπέδιο. Για παράδειγμα, εγκλήματα πολέμου. Και δεν μιλώ για επί αλλά τα πρόσωπα. Με τον Herbert Bush το 2009 είχαμε επισκεφθεί τον ΟΗΕ διότι ο ΟΗΕ δεν είχε ε, υλοποιήσει καμία ε, από τις, ε, ε, από τις εντολές συλλήψεων που είχαν εκδοθεί. Ο κ. Ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που είπατε για τη διάρκεια των ερευνών και τα διαδικαστικά δικαιώματα. Όμως ε, σημαντικό είναι και για αυτόν που κάνει την έρευνα να ολοκληρώνεται γρήγορα η έρευνα. Αυτό αφορά και τα κρατημέλη, τι ε, τις υποθέσεις δηλαδή για τις οποίες ήταν αρμόδιος ενώπιον των κρατομελών, αλλά και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζετε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό ή η έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνονται εξωτερικά. Και ποιο είναι ο ρόλος τη εποπτική επιτροπή ε, με βάση και τις ε, ε, τριβές που υπήρξαν στο παρελθόν, πώ ακριβώς θα, θα τις αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, δικονομικά δικαιώματα, ελεγκτές ε, και Εποπτική Επιτροπή. Αυτά τα τρία ερωτήματά μου. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικά αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε. Αρχικά, διερευνητικά ε, δικαιώματα και τα δικαιώματα του, του εμπλεκόμενου θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη, γιατί εκεί είναι το βασικό μέλημα. Ε, εκεί γίνεται η ανάλυση των δεδομένων, εκεί ε, στοιχειοθετείται η υπόθεση. Όλα αυτά απαιτούν στήριξη και από ισχυρή εύρωστη εξωτερική επαλήθευση. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με, την, με το ρόλο της Εποπτικής Επιτροπής. Δεν έχουμε εμπειρία ακόμα για τα διαδικαστικά δικαιώματα, γιατί ακόμα, δεν έχουν προσδιοριστεί. Αλλά έχω, είναι ένα προτέρημά μου αυτό ένας τομέας ειδικότητας, η λειτουργία εντός δικτύων. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα δικαιώματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με, τη διερεύνηση. Αντιθέτως, καμία σωστή έρευνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς σεβασμό στα δικαιώματα του ερευνομένου. Επομένως πρέπει να έχουμε και τις δύο υποθέσεις, και εξωτερικό και εσωτερικός έλεγχο. Ένα ερώτημα, ποια είναι η γνώμη σας, λέει ο κ. Βάλλη, ε, οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αρκετά για την καταπολέμηση ε, αυτή τη μάστιγα σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και απονομική ε, σκοπιά ε, κτλ. Ευχαριστώ. Το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται ακριβώ στο επίκεντρο αυτή τη μάστιγα ε, που στερεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα στο παρελθόν, και αυτό και είναι γεγονό αυτό, είχε κάποιε εισαγγελικέ αρμοδιότητε, αλλά δεν ήταν πραγματικά εισαγγελική αρχή και γι' αυτό δεν είχε δυνατότητα να το αντιμετωπίσει. Γιατί ό,τι στοιχεία και να παρουσίαζε ο Όλαφ δεν αντιμετωπιζόταν ω ε, στοιχείο από τα κράτη-μέλη. Η λειτουργία λοιπόν, η θέσπιση τη εισαγγελία είναι, είναι πραγματικό βήμα προόδου, γιατί κλείνει αυτό το κενό. Για το οργανωμένο έγκλημα βλέπουμε ότι αναφέρεται και στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην οδηγία PIF και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν πετύχει, και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πετύχει, ε, θα αξιοποιήσει στο έπακρο και το τελευταίο ευρώ και θα βελτιώσει ε, τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί συνήθω γίνεται διασυνοριακά αυτή η εγκληματική δραστηριότητα με μεγάλα ποσά και δεν μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς τη συνεργασία των εθνικών ε, δικαστικών αρχών. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα θα πρέπει ε, να απενδυθεί αυτές τις ε, ήμοι εισαγγελικέ αρμοδιότητες και να συνεργαστεί και με τις εθνικές αρχές, ε, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί υπάρχει διαφορετική μεταχείριση προσώπων που είναι ερευνόμενα ανάλογα ε, εάν συμμετέχουν στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι ή που δεν θα προσχωρήσουν στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν θα ευαισθητοποιήσει τις έρευνες, δεν αποτελεί αρνητικό πρόκριμα, διότι μιλάμε για το δικαίωμα υπεράσπισης αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολίτες ερευνόμενοι που θα έχουν αυτές τις εγγύησεις, ενώ σε μια παρόμοια υπόθεση άλλοι πολίτες δεν θα έχουν τις ε, ίδιες εγγύησεις γιατί προέρχονται από μια χώρα που δεν ε, έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν θα αποσαφρώσει κάπως ε, την όλη διαδικασία έρευνας απάντηση. Πολύ δύσκολη η ερώτηση γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορεί ο Γενικός Διευθυντής του Όλαφ να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ μαζί σας ότι Υπάρχει opt-in και opt-out χωρών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν θέλω να είμαι κοινικός, θα μπορούσα να πω ότι το ναι, στην περίπτωση του ναι, οι έρευνες θα παραμείνουν στα πλαίσια του Όλαφ. Δεν σκέφτομαι όμως έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι τα καλά αποτελέσματα και τα πιστικά στοιχεία που θα δώσει η Ευρωπαϊκή η Εισαγγελία έτσι ώστε να δράσει ως μαγνήτης και να προσχωρήσουν και οι χώρες που θα δουν τα καλά αποτελέσματα και την ομοιογένεια αποτελεσμάτων, να φτάσουμε σε μία εναρμόνιση ε, αντίντεριμ μπορώ να πω ότι ο Όλαφ ε, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι προδιαγραφές του Όλαφ να είναι οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον σε παρόμοιες υποθέσεις. έτσι ώστε, όπως είπατε και εσείς, να αποφύγουμε κάθε σκιά. Νόβακοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μίλσκε, ζούμε σε καιρούς ε, εγγράφων του Παναμά, ε, Paradise Papers, ό,τι έγγραφα θέλετε. Ζούμε σε ε, καιρούς κοινοπραξιών όπου μια εταιρεία ανήκει σε μια άλλη υπεράκτεια η οποία ε, υπάγεται σε χι άλλες υπεράκτειες έτσι ώστε να μην ελέγχονται οι τραπεζικοί οργανισμοί, ε, συγγνώμη, λογαριασμοί πλήρως. Θεωρείτε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις διότι ο ο Όλαφ μαζί με αυτή την Επιτροπή είναι ο καλύτερος φίλος του φορολογούμενου. Απάντηση. Συμφωνώ ότι εμείς και εσείς, ε, μάλλον ο Όλαφ και εσείς, είσαστε, είμαστε, είσαστε οι καλύτεροι φίλοι του φορολογούμενου. Πρόσβαση τώρα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ξέρω ότι αναφέρεται το θέμα στις εκθέσεις του Όλαφ. Αποτελεί μία πρόκληση. Θα πρέπει να δούμε την όλη διαδικασία, το όλο ταξίδι αυτό και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε τις ε, πληροφορίες, όπως είπατε. Ο δημόσιος κατήγορος λοιπόν θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να προβεί σε εθνικές δικαστικές διώξεις και ο Όλαφ θα συνδράμει. Δεν θα συνέδραμα εάν ο Όλαφ έκανε δικές του έρευνες και διώξεις εκτός Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα για την απάτη στον ΦΠΑ όπου θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ ε, κρατών μελών και Όλαφ ε, χρήζει βελτιώσεων, ιδίως και με βάση τις γερμανικές απόψεις για τις αρμοδιότητες του Όλαφ. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιωθεί η συνεργασία σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, η αρμοδιότητα για υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ παραμένει στον, ε, για τη διερεύνηση των υποθέσεων ε, παραμένει στον Όλαφ εφόσον οι υποθέσεις αυτές δεν είναι διασυνοριακές και δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό. Συνεργασία. Θεωρώ ότι είναι σημαντική αλλά όχι μόνο στον τομέα των ερευνών. Η διερεύνηση μιας απάτης ακολουθεί πάντοτε τα χρήματα, γιατί τα χρήματα ε, πάντοτε ε, φέρνουν απάτη. Ε, οι απάτες πάντοτε συγκεντρώνονται εκεί που υπάρχουν τα πολλά χρήματα. Η απάντηση που και η λύση για, να, για αυτό το πρόβλημα είναι η εναρμόνιση των δικαιικών συστημάτων και την καταπολέμηση κενών και παραθυρακίων που υπάρχουν στην νομοθεσία, γιατί αυτά αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται οι απαταιώνες. Ο Όλαφ λοιπόν, κατά την δική μου θεώρηση, πρέπει πάντοτε να είναι σημαντικός εταίρος στο πλαίσιο της νομοθεσίας προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες να προβεί σε, σε απάτη. Και αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζω στεναρά. Και εγώ να ρωτήσω εκ μέρους του ΕΛΚ ποια είναι η άποψή σας για τις διαδικασίες ε, clearing house, γραφείων συμψηφισμού. Εκεί όπου συναντάται ο διευθυντής του Όλαφ με τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσει θέματα που αφορούν το προσωπικό της Κομισιόν. Τι, πώς πιστεύετε ότι εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του Όλαφ σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, κατάλαβα την υπόθεση του Κωσόβου, αλλά έχουν παρέλθει από τότε 15, 16, 17 χρόνια. Ποιες είναι οι εμπειρίες σας στον τομέα των ε, αστυνομικών ερευνών. Ευχαριστώ. Πρώτον, για τα γραφεία συμψηφισμού. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι ο Γενικός Διευθυντής του Όλαφ ε, ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα όταν ερευνώνται ε, πρόσωπα, μέλη του προσωπικού ε, της Κομισιόν. Γνώμη μου είναι ότι εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί έρευνες, ΟΛΑΦ πρέπει να έχει πλήρη ερευνητική ανεξαρτησία. Καταλαβαίνω ε, τη θέση του Όλαφ στο οργανόγραμμα της ε, Κομισιόν. Ε, το έχω μελετήσει σε βάθος και καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε μπορεί να έχει επιπτώσεις. Εγώ προσωπικά όμως ποτέ, ποτέ δεν έχω παζαρεύσει και δεν έχω επιδοθεί σε συζητήσεις πριν από την ολοκλήρωση ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία 25 χρόνια. Ε, πολύ πρόσφατα έχω αποκτήσει εμπειρία ε, όσον αφορά τη συνεργασία με αστυνομικέ αρχές και θα πω ότι ε, ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή ε, είναι συμμόρφωση, αφορά τη συμμόρφωση με κώδικες διεντολογίας και αυτό είναι σημαντικό γιατί θεωρώ ότι ο Όλαφ πρέπει να καταστεί και ε, φορές διαχείρισης κινδύνου. Τα τελευταία δέκα χρόνια από τη θέση μου έχουμε συλλέξει πληροφορίες, έχουμε φέρει υποθέσεις ε, σε, στη δικαιοσύνη σε χώρες και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μάλιστα ακόμη και σε χώρες όπου τα δικαιικά συστήματα, τα συστήματα της δικαιοσύνης είναι πολύ αδύναμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν στέφτηκαν όλες οι προσπάθειές μας με, ε, ε, με απόλυτη αποτυχία. Κάποιες ε, δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν, κάποιες από τις έρευνές μας δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν ήρθα εδώ για να σας πω τι τέλειος που είμαι, αλλά να σας παρουσιάσω το έργο μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε βεβαίως για την παρουσία σας και ε, θα συνεχίσουμε εμείς θα δώσω τώρα πέντε λεπτά στις ε, πολιτικές ομάδες προκειμένου να γίνει η εσωτερική συζήτηση και στη συνέχεια θα ε, προχωρήσουμε στην υποφορία. Πέντε λεπτά διάλειμμα.